Goedemorgen iedereen. We hervatten eh, de vergadering die... Eh, Καλημέρα, επαναλαμβάνω τη συνεδρίαση που είχε διακοπεί χτες και περνάμε κατευθείαν στις ε, ψηφοφορίες, στην ψηφοφορία της ε, έκθεσης της κυρίας Μακοβέη, το σημείο 11. Είναι εδώ πέρα η συγγήτρια. Κυρία Μακοβέη, θέλετε να πείτε κάτι. Καλημέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, τους χειώδεις συγητές με τους οποίους είχα πολύ καλή συνεργασία. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ναι. Ε, σας ευχαριστώ. Πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι τεχνικό. Είναι στην ε, στον κατάλογο, αλλά θέλω να γραφτεί στα πρακτικά. Εκεί πέρα που λέγεται Μακεδονία πρέπει να αντικατασταθεί με το Πουγουδουμού. Αυτό είναι η σωστή διατύπωση. Μάλιστα το σημειώσαμε. Ξεκινάμε με την ε, ψηφοφορία. Λάθος κατάλογο έχω εγώ. Ναι. Άφετ 1 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Άφετ 2 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 10 της κυρίας Μακοβέη με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Παράγραφος 2, πίνακας 1, προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 11 χαρτόγκο υπέρ. Κατά. Αποχές. δε, Απορρίπτεται. 12 επίσης χαρτόγκο υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 4 πίνακας 2 Μακοβέη και Κάλβιν υπέρ κατά αποχές δεκτή 13 χάρτον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 Μακοβέη υπέρ κατά αποχές δεκτή 15 Μίλντερ υπέρ κατά αποχές δεκτή 16 17 και 18 καλύπτονται από μια συμβαστική υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Γίνεται δεκτή, οπότε η παριθμό 19 καταπίπτει. Παράγραφος 6, πίνακα 3, Μακοβέ και Κάλπιν υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 20 Κάλβιν καλύπτεται από το συμβαστική 3, οπότε δεν χρειάζεται να ψηφιστεί. Μετά 21, 22, 23, 24 καλύπτονται από τη συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ο Κριστιαν μου λέει εδώ πέρα πως Παρά το ότι έγινε δεκτή η συμβαστική 3 πρέπει να ψηφίσουμε την υπαριθμόν 22 της κυρίας Μακοβέ υπέρ κατά αποχές δεκτή περνάμε στην ΑΦΕΤ 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 25 χάρτο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 27 πακοβέει υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 28 μακοβέει υπέρ κατά αποχές να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά την 28 της κυρίας Μακοβέη. άρχη ψηφοφορία. Έχετε 5 δευτερόλεπτα κύριε Γεκαΐρ. Ωραία. Πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτή 16 εναντί 6. 29 Μακοβέη υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Παράγραφος 8 Δέλτα. Νέα παράγραφος, προφορική τροπολογία επίσης κυρίες Μακοβέ υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Άφετ 7 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 30, 31, 32 καλύπτονται αυτές από τη συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή αφέτ 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 33 της κυρίας Μακοβέ υπέρ κατά αποχές δεκτή 34 της κυρίας Μακοβέ υπέρ κατά αποχές δεκτή 35 Μακοβέ υπέρ κατά αποχές δεκτή 36 της κυρίας Μακοβέ υπέρ κατά αποχές δεκτή 37 του κυρίου Χάρτον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 Κάλβιν υπέρ κατά αποχές δεκτή 39 δικιά μου υπέρ κατά αποχές δεκτή άφετ 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή άφετ 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 40 μακοβέ υπέρ κατά αποχές δεκτή 41 δική μου και της κυρίας Μακοβέ υπέρ κατά αποχές δεκτή 42 χάρτον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 μακοβέι υπέρ κατά αποχές δεκτή περνάμε στην 44 προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή 45, 46, 47 καλύπτονται από τη συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 48 χάρτονγκ καταπίπτει 49 της κυρίας Μακοβέη υπέρ κατά αποχές δεκτή 50 χάρτονγκ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 Μακοβέη υπέρ κατά αποχές δεκτή 52 Μακοβέ. υπέρ κατά αποχές δεκτή 53 χάρτον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 μακοβέ υπέρ κατά αποχές δεκτή 55 κάλφιν όχι 54 ναι, έχει γίνει δεκτή, οπότε 55 καταπίπτει, 56 Μίλτερ υπέρ. Κατά, αποχές δεκτή, 58 Κάλφιν υπέρ. Κατά, αποχές δεκτή, 57 είναι συμβατή με την 58, 57 υπέρ. Κατά, αποχές δεκτή, 59 υπέρ. Κατά, αποχές δεκτή, 60 Μακοβέη υπέρ κατά αποχές δεκτή 61 Μακοβέη υπέρ κατά αποχές δεκτή 62 Μάλετιτς υπέρ κατά αποχές νομίζω πως απορρίπτεται θα το επαληθεύσουμε 62 Μάλετιτς Πέρας. Πράγματι απορρίπτεται. Ε, δεν σηκώνετε τα χέρια σας όμως. Λίγο πιο ενεργητικά την άλλη φορά. Λοιπόν, 63. στάσμα κοβέ υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 64. μακοβέ υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 65. μακοβέ υπέρ κατά αποχές δεκτή 66 Κάλβιν αποσύρεται 67 Μάλετη Τσιπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 Μακοβέη 68 μέχρι και όχι πρέπει μία μία Καλώς. 68 Μακοβέη υπέρ κατά αποχές δεκτή 69 Μακοβέ υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 74 υπέρ κατά αποχές δεκτή 75 υπέρ κατά αποχές δεκτή 76 υπέρ κατά αποχές Μ, δεν είμαι σίγουρος 76 λοιπόν να την επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά δεκτεί Δεκτή. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτό δεν είναι σαφές. Να επαληθεύσουμε και την 77 της κυρίας Μακοβέη. άρχιε την ψηφοφορία. Πέρας. 13-11. Μάλιστα. Δεκτή. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πως είναι η ίδια πάλι πλειοψηφία, αλλά θα... Α, εντάξει, δεκτή. Συμφωνείτε? 79 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 81 υπέρ κατά εποχές δεκτή 82 υπέρ κατά αποχές δεκτή 83 υπέρ κατά αποχές δεκτή 84 υπέρ κατά αποχές δεκτή 85 υπέρ κατά αποχές δεκτή 86 υπέρ κατά αποχές δεχτεί 87 υπέρ κατά αποχές δεχτεί 88 υπέρ κατά αποχές δεχτεί 89 υπέρ κατά αποχές δεχτεί 90 υπέρ κατά αποχές δεχτεί 91 υπέρ κατά αποχές δεκτή 92 υπέρ κατά αποχές δεκτή 93 υπέρ κατά αποχές δεκτή 94 υπέρ κατά αποχές δεκτή 95 υπέρ κατά αποχές δεκτή 96 κάλφιν πίπτη γιατί πέρασε 95. Περνάμε στις ιδεολογικές σκέψεις. Τροπολογία 1, Γιάν Μίλτερ, προφορική τροπολογία, υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτή. Α, ήταν σε μέρη. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος. Μέρος δεύτερο, υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτή. Μέρος τρίτο καλύπτεται από τη συμβαστική 1 Ψηφίζουμε τώρα τη συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Μέρος τέταρτο καλύπτει από τη συμβαστική 2. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Μέρος 5 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 2 του κυρίου Χάρτονγκ καταπίπτει γιατί έχει γίνει δεκτή 1 και περνάμε στις 3 ε, και 4 Α, καλύπτονται οπότε έχουν ήδη ψηφιστεί με τη συμβαστική 1 τροπολογία 5 μακοβέη υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 6 και 7 καλύπτονται από τη συμβαστική 2 δεν χρειάζεται λοιπόν να ψηφίσουμε τροπολογία 8 Κάλφιν υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 9 Μακοβέη υπέρ κατά αποχές δεκτή περνάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία που ούτως ή άλλως θα γίνει ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρας ομόφωνα. Συγχαρητήρια κυρία Μακοβέη. Περνάμε στην έκθεση της κυρίας Τσέσκοβα. Με ακούσατε. Να έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. η διαδικασία απαλλαγή για το Συμβούλιο και για πρώτη φορά εφέτος και για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για πρώτη φορά είναι ένα είδος ετήσιας μάχης που δίδεται μεταξύ Κοινοβουλίου και ε, του Συμβουλίου σε σχέση με το ποιο από τα δύο αυτά όργανα έχει μεγαλύτερες αρμοδιότητες για τη διαδικασία απαλλαγής. Δυστυχώς. Το ίδιο πράγμα είναι και το 2011. Είναι η δεύτερη φορά που μας απασχολεί το θέμα αυτό εδώ. Πιστεύω ότι πέραν του θέματος των αρμοδιοτήτων και των διαφορετικών νομικών νορμοδοτήσεων που μας έχουν υποβληθεί, πιστεύω ότι αν δεν απαντηθούν όλα τα ερωτήματα τα οποία έχει θέσει το Κοινοβούλιο, θα πρέπει να είμαστε συνεπείς με τον εαυτό μας και θα πρέπει όπως και τα προηγούμενα χρόνια να πράξουμε <clears throat> και πιστεύω ότι δεν μπορούμε να αποφασίσουμε διαφορετικά εφέτος, θα πρέπει και εφέτος να απορρίψουμε την ε, <clears throat> απαλλαγή, να μην δεχτούμε την απαλλαγή. Αυτό είναι το περιεχόμενο της δεύτερης έκθεσής μου. Η ελπίδα μου είναι ότι στο μέλλον κάποιος διαφορετικός εισηγητής θα μπορέσει να βρει μια καλύτερη λύση θα ήθελα πάρα πολύ το Συμβούλιο να μπορούσε να αναπτύξει ένα πιο επικοδομητικό διάλογο μαζί μας, με τα μέλη της Επιτροπής μας. Όπως έχουν όμως τώρα τα πράγματα, το μόνο που μπορώ να προτείνω είναι αυτό το οποίο έχω στην εκθεσή μου και ζητώ και οι συναδελφοί μου να υποστηρίξουν την εκθεσή μου για την απόρριψη της απαλλαγής. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να απαντήσει εξ ονόματος του Συμβουλίου. Βλέπω πως απουσιάζει το Συμβούλιο, αλλά μια που οπωσδήποτε μας βλέπουν από το ίντερνετ, θα δουν πως θα ψηφίσουμε. Υπάρχει κάποιος άλλος να που θέλει να πει κάτι. Όχι. Περνάμε στην ψηφοφορία. Πρώτη πρόταση για απόφαση, παράγραφος 1, τροπολογία 1 του κυρίου Οντή, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2 σόντερ υπέρ κατά αποχές δεκτή μετά ψηφίζουμε την πρόταση απόφασης όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά και η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 23-1. περνάμε στο ψήφισμα παράγραφος 9 τροπολογία 3 τσέσκοβα υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 4 τσέσκοβα υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 5 σόντερκάρτ υπέρ κατά αποχές Νομίζω πως απορρίπτεται. Ε, την επαληθεύσουμε όμως. 5 Sondergaard, ηλεκτρονικά. Πέρας. 13 11 γίνεται δεκτή. 6 Τσέσκοβα καταπίπτει. Τροπολογία 7 Sondergaard. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 8 Σόντεργαρντ υπέρ κατά αποχές δεκτή τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική άρχεται η ψηφοφορία πέρας ομόφωνα εγκρίνεται συγχαρητήρια κυρία Τσέσκοβα Ωραία. Τελείωσαν οι ψηφοφορίες. Και... Ε, μπήκαν όλοι στην αίθουσα. Επισκέπτες και collega's, ik ga eventjes moeten eh, pauzeren, want... Κάνουμε ένα διαλυματάκι, συνάδελφοι, γιατί το θέμα για την ε, έκθεση σχετικά με την προστασία των οικονομικών σφαιρότων της Ένωσης και καταπολέμηση της απάτης ε, της κυρίας ε, Γιάλα Σέντερ δεν ξέρω αν μπορεί να συζητηθεί χωρίς τον κύριο Σεμέτα και τον κύριο Κέσλερ Οπότε θα τους περιμένουμε και αναβάλλεται, διακόπτε με συγχωρείτε για λίγα λεπτά η συνεδρίαση. το από Goed, collega's. We gaan de Συνεχίζεται η συνεδρίαση, συνάδελφοι. Πάμε στο σημείο 13. Συζήτηση δύο εκθέσεων. Τελικά, έκθεση για την προστασία των οικονομικών σφαιρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα το παρουσιάσει ο κύριος Σεμέτα και την έκθεση του Όλαφ που θα την παρουσιάσει ο κύριος Κέσλερ. Προτείνουμε να κάνει μια πρώτη εισαγωγή ο κύριος Σεμέτα, η κυρία Σέντερ, η συγγήτρια, να απαντήσει, να συζητήσουμε και μόλις τελειώσουμε με αυτό θα ακούσουμε τον κύριο Κέσλερ και μετά ε, η κυρία Σέντερ και συζήτηση. Συμφωνείτε, δύο πράγματα ακόμα. Εγώ πρέπει να φύγω στις 10 η ώρα γιατί είμαι σε άλλη επιτροπή συγητής ε, για την ε, αποστολή παράνομων αποβλήτων και θα με αντικαταστήσει ο κύριος Λιμπεράτσικη από τις 10 ώρα και δεύτερον δύο και μισή υπάρχει συνέντευξη τύπου για την επίσκεψη της αντιπροσωπείας ε, στην Βουλγαρία και στο Καλίνιγκραντ και καλό είναι να είναι παρόντες όσοι πήγαν στην αίθουσα ASP 5K3 στην αίθουσα τύπου. Κύριε Επίτροπε, έχετε τώρα τον λόγο για να μας ε, παρουσιάσετε την έκθεση. I am pleased to present to you the Commission's 2012 annual report on the protection. Με χαρά σας παρουσιάζω την ετήσια έκθεση της Κομισιόν του 2012 για την προστασία των, των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προστασία από απάτες. Είναι ένα βασικό στοιχείο της προσπάθειας διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πώς γίνεται η διαχείριση και ο έλεγχος των κονδυλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο μας επιτρέπει μια γενική επισκόπηση κατάσταση σε κάθε κράτος μέλος, αλλά επίσης μας βοηθάει να, να εντοπίσουμε συγγνώμη, τα σημεία αδυναμίας. Μας επιτρέπει έτσι να έχουμε κάποιο στόχο θετημένες δράσεις κατά των απατών και των ατασταλιών. Η έκθεση δίνει μια επισκόπηση όλων των ατασταλιών που έχουν αναφερθεί στην Κομισιόν από τα Κάτι μελη το 2012 και επίσης των μέτρων που ελήφθησαν για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Περιλαμβάνει επίσης και συστάσεις για μελλοντική βελτίωση. Η μέθοδος παροχής αναφοράς ε, χρησιμοποιεί και δύο πρακτικές που εισήχθησαν πες και που θεωρούνται πολύ χρήσιμες. <clears throat> Μια σαφή διάκριση μεταξύ ε, ατασταλιών που έχουν χαρακτήρα απάτης και αυτών που δεν είναι απάτης και δεύτερον η πρακτική εναρμόνιση των πληροφοριών για τα προληπτικά και τα επανορθωτικά μέτρα βάσει των στοιχείων που βρίσκονται στους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τω μεταξύ υπάρχουν δύο σημαντικά νέα στοιχεία στην ετήσια έκθεση του 2012 που αντανακλούν και σχόλια της δικής σας Επιτροπής σε σχέση με προηγούμενες εκθέσεις. Πρώτον, έχουμε ενισχύσει την ε, σύνδεση μεταξύ της, ε, του εντοπισμού και της αναφοράς των στοιχείων αυτών από τις εθνικές αρχές. Είμαστε πεπισμένοι ότι έχει βελτιωθεί σημαντικά η αναφορά τασταλιών έναντι των προηγουμένων ετών. Είναι μια πρόοδος αυτό ήδη. Όπως θυμόσαστε, τα προηγούμενα χρόνια είχα εκφράσει ανησυχίες ότι η ίδια η ποιότητα των αναφορών δεν ήταν επαρκής. Εάν όμως θεωρήσουμε τώρα ότι οι απάτες οι οποίες ανακαλύπτονται αναφέρονται τώρα τις περισσότερες φορές στα έγγραφα των κατών μελών, θα πρέπει να δούμε και τα στοιχεία. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα για τις χώρες αυτές που είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο της απάτης που αναφέρεται. Ο μικρός αυτός αριθμός ατασταλιών που αναφέρεται δείχνει πράγματι ότι είναι κοντά στο μηδέν το ποσοστό απάτης στις χώρες αυτές ή σημαίνει ότι υπάρχουν προβλήματα με τον εντοπισμό της απάτης στις χώρες αυτές. Αυτό είναι ένα θέμα που θα το ερευνήσει ενδελεχώς η Κομισιόν. Το δεύτερο νέο στοιχείο στην έκθεση του 2012 είναι μια ευρύτερη ανάλυση αυτών των ατασταλιών που έχουν παρουσιαστεί ως απάτες από τα κράτη-μέλη για να δούμε ποια είναι η φύση τους και ποιος είναι ο τρόπος αντιμετώπισης τους στα κράτη-μέλη. Τέλος, σε επίπεδο δομής. Η έκθεση, όπως πάντα, περιλαμβάνει και πρόσθετες πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εστιάσαμε στους ελέγχους στον τομέα της γεωργίας. Υπάρχουν παρατήματα, λοιπόν, ε, στην έκθεση που δίνουν και μια επισκόψη του προγράμματος Ηρακλής 2. Τώρα, αν σταθούμε στα αριθμητικά στοιχεία, βλέπουμε ότι ο συνολικός αριθμός των, ε, ε, απατών 1231 με ύψος 930 εκατομμύρια ευρώ έχει παραμείνει γενικά σταθερός εναντί του 2011. Αλλά υπάρχει μια αύξηση κατά 8% σε ό,τι αφορά τις απάτες στον τομέα δαπανών, αυτό συνδέεται σχεδόν απόλυτα σε δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις για προενταξιακά κονδύλια που βρίσκονται τώρα ενώπιον στη δικαιοσύνη στις αντίστοιχες χώρες. <clears throat> σε ό,τι αφορά τις, τα έσοδα, έχουν μειωθεί κατά 30% περίπου οι απάτες έναντι <clears throat> του προηγούμενου έτους και πρόκειται για 77 εκατομμύρια ευρώ άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες σε σχέση με τους τομείς όπου γίνονται οι απάτες, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι υποθέσεις αυτές, όλα αυτά αναφέρονται στην έκθεση. Οι ατασταλίες που δεν έχουν χαρακτήρα απάτης και ο αντίκτυπός τους, ο οικονομικός, ήταν πιο μεγάλος το 2012. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι εφαρμόστηκαν δημοσιονομικές <clears throat> ε, διορθώσεις όταν έκλεισε το, το πρόγραμμα για την πολιτική συνοχή. Επίσης, προγράμματα που συνεχίζονται έχουν, ε, εντατικό, ε, έχουν εφαρμοστεί πιο εντατικά γιατί τελειώνει η ε, περίοδος προγραμματισμού. Είναι επίσης σημαντικό ότι η Κομισιόν ανέκτησε ή διόρθωσε 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ αχρεωστήτως καταβληθέντα πέρσι. Και πήραμε και 187 αποφάσεις για να διακόψουμε πληρωμές ύψους 5 δισεκατομμύριων ευρώ στην πολιτική συνοχής. Και <clears throat> υπήρξαν τέσσερις αποφάσεις αναστολής που εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι το τέλος του 2012. Όλα αυτά δείχνουν ότι οι μηχανισμοί αυτή προστασίας του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χρημάτων των φορολογουμένων μας λειτουργούν αποτελεσματικά. Περνάω σε ένα άλλο σημαντικό συμπέρασμα που μπορούμε να αντιλήσουμε από την έκθεση του 2012. Οι αναφορές για τις απάτες φαίνεται ότι έχουν βελτιωθεί συλλήβδιν, αλλά υπάρχουν ακόμα αποκλίνουσες προσεγγίσεις για την ε, εντοπισμό και τη συνέχεια που δίδεται στις απάτες αυτές. Κάποια κρατημέλη αποδίδουν σημαντικούς πόρους στην καταπολέμηση της ε, απάτης, αλλά κάνουν απλώς δημοσιονομικές προσαρμογές χωρίς να ψάχνουν περισσότερο δυνητικά εγκληματικές ενέργειες. Όπως βλέπουμε υπάρχει διαφορά όχι μονάχα μεταξύ κρατών μελών, αλλά και μεταξύ διαφορετικών διοικητικών αρχών στην ίδια χώρα. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό, <clears throat> δεδομένου του ότι ως μια ένωση με ενιαία αγορά και κοινό προϋπολογισμό είμαστε τόσο ισχυρή όσο ο ασθενέστερος μας κρίκος σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της απάτης. Αυτό όμως πάλι δεν μας εκπλήτηκε τόσο πολύ. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η Κομισιόν έκανε συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες που θα σας αναφέρω σε λίγο. Πιο θετικά μπορώ να σας πω ότι οι ορισμένε δράσεις οι οποίες είχαν αναλυθεί για να βελτιωθεί η προστασία του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχίζουν να έχουν πραγματικό αποτέλεσμα. Παραδείγματος χάρη υπάρχει μια σαφή στάση που αναφέρεται στην έκθεση ότι οι μισές από τις ε, απάτες α, έχουν εντοπιστεί από εθνικές ή ευρωπαϊκές αρχές και επίσης κατά τη διάρκεια ποινικών ερευνών. Τα οι άλλες μισές όμως βρέθηκαν με διοικητικούς ελέγχους που προβλέπονται από, τις κατατομή. ε, από τους κατατομής κανονισμούς. Αυτό είναι καινοφανές και επικυρώνει την απόφασή μας που αναφέρθηκε στην έκθεση του 2001 να έχουμε πιο δομημένη συνεργασία όλων των υπευθύνων για τη διαχείριση των κονδυλίων. Βλέπουμε ότι τα κάτι μελη έχουν δώσει συνέχεια σε πολλές συστάσεις που τους έγιναν στην έκθεση του 2011. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη χρήση του συστήματος IRMS και των εθνικών στρατηγικών για τα, για τα ε, δασμολογικά έσοδα. Να σας κάνω τώρα μια σύνομη επισκόπηση των κυρίων πολιτικών κατά της απάτης που έχει ξεκινήσει η πολιτική τα τελευταία χρόνια. Περιλαμβάνεται πρώτα την εφαρμογή μιας νέας αντιαπατηλής στρατηγικής, την οποία ανέφερα προηγουμένως. Παραγωγός χάρη, ρήτρες κατά των απατών έχουν συμπεριληφθεί σε πολλές διεθνείς συμφωνίες συνεργασίας και στις προτάσεις της Κομισιόν για νέους ε, κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες. Τον Ιούλιο του 2012 μαζί με την Επίτροπο και αντιπρόεδρο κυρία Ρέντινγκ παρουσιάσαμε μια πρόταση οδηγία για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τη χρήση του ποινικού δικαίου. Ο στόχο τη πρόταση αυτή είναι να εξασφαλίσουμε μια πιο εναρμονισμένη προσέγγιση στον κολασμό των αδικημάτων κατά του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι εγκληματίε να μην εκμεταλλεύονται τι διαφορέ μεταξύ των εθνικών νομικών συστημάτων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για να εξασφαλίσει ότι αυτή η νομοθεσία θα εφαρμοστεί ορθά. Θα επανέλθω όμω ως ο νούπος στο θέμα αυτό. Τον Ιούλιο του 2012 παρουσιάσαμε μια α, φιλόδοξη πρόταση για ένα ευρωπαϊκό εισαγγελικό γραφείο. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε έναν εξάρτητο φορέα ο οποίος θα δώσει πρώτη προτεραιότητα στον αγώνα κατά της απάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αυξήσει την επιτυχία των προσπαθειών μας. Μαζί με την πρόταση αυτή για την εισαγγελική αρχή υπήρχε και μια ανακοίνωση για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε καλύτερα την διακυβέρνηση της όλα. Εγώ προσβλέπω σε μια σε βάθος συζήτηση μαζί σας τους επόμενους μήνες σε σχέση με αυτή την πρωτοβουλία και θα ήθελα να ακούσω και τις δικές σας απόψεις για όλες αυτές τις ιδέες που έχουμε εμείς παρουσιάσει. Έντιμα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Η έκθεση του 2012 μας υπενθυμίζει ότι ενώ έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπίσουμε την απάτη προς τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλής δρόμος παραμένει για να τον διατρέξουμε. Πολλά κράτη-μέλη έχουν δώσει μια σχετικά χαμηλή προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των απατών προς τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εθνικές απόψεις αποκλίνουν και διαφέρουν σημαντικά. Οι προτάσει που έχουν υποβληθεί από την Κομισιόν για το, την Εισαγγελική Αρχή θα εξασφαλίσουν ότι οι απάτες θα τύχουν της πρέπουσας προσοχής και αντιμετώπισης όπου και να λαμβάνουν χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ως εκ τούτου ότι αυτές οι σημαντικές πρωτοβουλίες θα μπορούν να υλοποιηθούν ως νομοθεσία το ταχύτερο δυνατό. Για την οδηγία TIF ξέρετε ότι η γενική <clears throat> ε, αντιμετώπιση του Συμβουλίου ήταν να αποδυναμώσει την πρόταση της Κομισιόν οι αλλαγές οι οποίες έγιναν από το Συμβούλιο ουσιαστικά απειλούν και το υπάρχον και εκτιμένο. Έρχομαι εδώ για να ζητήσω από το Κοινοβούλιο λοιπόν να πάρει μια στεναρή θέση ε, υπέρ αποτελεσματικών κανόνων και να μην, ακολουθήσω τις, να μην ακολουθήσει τις απόψεις αυτές που θέλουν να μειώσουν το επίπεδο των ελέγχων για τον προϋπολογισμό. Ζητώ λοιπόν τη βοήθεια όλων των εντύμων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θέμα αυτό για να μας βοηθήσουν να καταλήξουμε σε μια αποτελεσματική προστασία του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Βασίζομαι και στη δική σας υποστήριξη για να εξασφαλίσω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή θα συμφωνηθεί και θα ε, υλοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό. Γιατί στο τέλος της ημέρας Ξέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι απόλυτα προσιλειωμένο στην, προσπα... στην προάσπιση των χρημάτων των φορολογουμένων όσο και η Κομισιόν. Η συνδυασμένη μας προσπάθεια και αφοσίωση σε αυτό το στόχο μπορεί να φέρει καρπούς. Σας ευχαριστώ και είμαι έτοιμος να συμμετάσχω στη συζήτηση. Ε, Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Πριν δώσω τον λόγο στην κυρία Γιάλα Σέντερ να δω ποιος άλλος θέλει το λόγο. Μακοβέη ο κύριος Μιλντερ. Μακοβέη, Μιλντερ, ο κύριος Φέρμπερ και ο κύριος Λιμπεράτσκι. Η κυρία Σάντερ έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Σεμέτα για την παρουσίαση που μας έκανε, τις ετήσιας έκθεσης για το 2012 που περιλαμβάνει όχι μόνο τα γνωστά <clears throat> στοιχεία που ξέρουμε κάθε χρόνο, αλλά μας φέρνει και νέα στοιχεία που είναι ιδιαίτερα θετικά, που βέβαια δεν είναι στην αρμοδιότητα την άμεση της Επιτροπής μας, γιατί είναι νομοθετικές προτάσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν από το Κοινοβούλιο αλλά και για την οδηγία και για το θέμα της εισαγγελικής αρχής. Όλα αυτά τα έχουμε υποστηρίξει εμείς και έχουμε δείξει πολύ θετικό ενδιαφέρον. Και είναι σαφές ότι έχετε την πλήρη υποστήριξη και συνεργασία μας. Εκ νέου παρά τις ε, προόδους οι οποίες επετέθησαν, βλέπουμε ότι όπως είπα, παρά το, τα θετικά στοιχεία από τον θετικό διάλογο μεταξύ των θετικών οργάνων, θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπουμε ότι παρά όλες αυτές τις βελτιώσεις που έχουν γίνει σε ό,τι αφορά τον αγώνα κατά της απάτης και για την καλύτερη παρουσίαση όλων αυτών των πορισμάτων έναντι της κοινή γνώμης, και αυτό το λέω γιατί άλλες πράξεις ατασταλίας είναι έχουν δόλο και είναι απάτες, άλλες είναι άδολες και δεν είναι απάτες. Είναι καλό λοιπόν η κοινή γνώμη να μπορέσει να καταλάβει αυτή τη διαφορά και όλα αυτά θα μας επιτρέψουν να έχουμε μια πιο σοβαρή αντιμετώπιση από την κοινή γνώμη και τους δημοσιογράφους. <clears throat> όλα αυτά λοιπόν είναι σημαντικά γιατί με τις ε, ε αλλαγές που έχουν γίνει το 2012 έχουν γίνει θετικές πρόοδοι. Βέβαια υπάρχουν και κάποια ερωτηματικά από τη μία πλευρά έχουν διατηρηθεί τα επίπεδα απάτη σε σχέση με το 2011. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν σημαντικές αυξήσεις σε ορισμένους τομείς. Μπορεί να είναι αποτέλεσμα της, ε, του, της περάτωσης προηγούμενης περίοδου δημοσιονομικού σχεδιασμού, αλλά μπορεί από την άλλη πλευρά να οφείλονται και σε άλλους παράγοντες, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες αυξήσεις στις απάτης που θα πρέπει να τις αναχαιτήσουμε. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε να είναι πιο χτυπητό <clears throat> είναι ότι από τη μία πλευρά και που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε λοιπόν είναι οι ελλείψεις οι οποίες παρουσιάζονται η έλλειψη μιας ομοιογενούς Κουλτούρα και κλίματος πολέμηση και πάταξη απάτης μεταξύ των κράτων μελών και φυσικά και μια ανομοιογένεια στον τρόπο που εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης της απάτης από τα κράτη-μέλη και έχουμε ένα ευρύ πεδίο δόξα σε ό,τι αφορά τη βελτίωση των μέτρων που εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη. Παραμένουν λοιπόν αυτές οι διαφορές όπως αναφέρατε προηγουμένως και η έκκληση που κάνετε για μια μεγαλύτερη ομοιογένεια και ενότητα των εργαλείων που χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη για μια κουλτούρα η οποία θα αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τις απάτες, αυτό δεν υπάρχει ακόμα. Θα ήταν πολύ χρήσιμο αυτό να υπάρχει βέβαια σε όλα τα κράτη-μέλη και σε όλες τις διοικητικές μονάδες οι οποίες αντιμετωπίσουν τη διαχείριση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δίωξη της απάτης. Είπατε ότι υπήρξε κάποια πρόοδος, υπήρξε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά παραμένουν σημαντικές διαφορές. Αυτό το οποίο εμένα με απασχολεί δεν είναι μονάχα αυτό που είπατε, οι διαφορές μεταξύ κρατών μελών, που μπορεί κανείς να το καταλάβει ότι είναι αποτέλεσμα διαφορετικής ιστορίας και κουλτούρας, αλλά και μέσα στα κρατη κράτη-μέλη τα ίδια υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ διοικητικών ε, δομών σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των ατασταλιών του προϋπολογισμού. Δηλαδή μέσα στην ίδια διοικητική μηχανή υπάρχουν διαφορετικές αντιμετωπίσεις. Προφανώς έχουμε να κάνουμε πάρα πολλή προσπάθεια και έχουμε ένα μακρύ και δύσκολο δρόμο για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το στόχο αυτό της ομοιογένειας που είπαμε προηγουμένως. Και είναι αλήθεια ότι τόσο η οδηγία όσο και το γραφείο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα θα βελτιώσουν την κατάσταση, αλλά μου φαίνεται πολύ σημαντικό, επειδή ακριβώς υπάρχουν αυτές οι διαφορές ε, μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ διοικητικών αρχών, και επειδή θα πρέπει να μεταγραφεί αυτή η οδηγία σε όλες τις χώρες μας και επίσης θα πρέπει να προστηρίσουμε καλύτερα την εντολή της εισαγγελικής αρχής, είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε κάποια ελάχιστα πρότυπα τα οποία να τηρούνται από όλα τα κρατημέλη σε σχέση με την καταπολέμηση της απάτης, αλλά να μπορέσουμε επίσης να εξασφαλίσουμε και μια δέσμευση όλων των κρατών μελών, ώστε να υπάρξει μια εναρμόνιση της κουλτούρας αυτής του αγώνα κατά της απάτης στο εσωτερικό των διοικητικών υπηρεσιών. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει ένα κεκτημένο σε επίπεδο ποινικού δικαίου ευρωπαϊκού για την καταπολέμηση της απάτης. Να μπορέσουμε έτσι με τον τρόπο αυτό να αποτρέψουμε τις ατασταλίες με μια καλύτερη γενική κουλτούρα, να ξεπεράσουμε την αδιαφορία για τον κοινωτικό προϋπολογισμό, να έχουμε καλύτερη εποπτεία και καλύτερο έλεγχο των ε, πληρωμών και των ε, συναλλαγών που συνδέονται με τον προϋπολογισμό να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις κινδύνου και να βελτιώσουμε την κατάσταση. Αυτά λοιπόν θα πω προς το παρόν, γιατί οι προτάσεις Κομισιόν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και φυσικά πρέπει να αντιμετωπιστούν από τον νομοθέτη. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να εργαστούμε λίγο περισσότερο στο να δούμε με ποιο τρόπο από τη βάση αυτής της έκθεσης που θα εκδώσει η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού μπορούμε να βοηθήσουμε την Κομισιόν στον δρόμο που έχει αναφέρει σε σχέση με την οδηγία και το, την, Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή για τις προτάσεις σε σχέση με την ΟΛΑΦ. Ήκοθ εννοείται ότι εγώ τις υποστηρίζω γιατί πρέπει να δοθούν περισσότερες εγγύησεις σε σχέση με την ΟΛΑΦ. Έχει τον κανονισμό της τον αυτόνομο, αλλά χρειάζεται να εστιάσουμε πολύ περισσότερο σε ορισμένε ε, πτυχές. Έχουμε δει βέβαια κάποια βελτίωση στις συζητήσεις που έχουμε κάνει προηγουμένω, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι πολιτέ μα θα καταλάβουν ότι είναι άσπυλο αυτό ο οργανισμό και δεν σκιάζεται από οποιαδήποτε αμφιβολία, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και φυσικά να εδραιώσουμε και την Ευρωπαϊκή Δυσαγγελική Αρχή. Όλα αυτά λοιπόν που έχει προτείνει η Κομισιόν είναι θετικά στοιχεία και τα οποία μπορούν να βελτιωθούν περισσότερο με τα σχόλια των συναδέλφων. Ευχαριστώ λοιπόν κύριε Επίτροπη και περιμένω τα σχόλια των συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αγιάλα Σέντερ. Κυρία Μακοβέη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Όπως γνωρίζετε το 2012 διαπιστώθηκαν πάνω από 1200 ατασταλίες πρόκειται για περιπτώσεις υποψίας ή ε, διαπιστωμένης απάτης και ε, το ποσό είναι σχεδόν 400 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περίπου όσο και την προηγούμενη χρονιά. Και το ερώτημά μου είναι το εξής. Αναφέρεται η εκτής έκθεση σε 9 υποθέσεις διαφθοράς σε τεσσερα κράτη-μέλη, Ιταλία, Κύπρος, Εστονία και Ισπανία, στον τομέα της πολιτικής συνοχής. Σε αυτές τις εννέα περιπτώσεις λοιπόν έχω τις ίδιες ερωτήσεις για τι είδους ε, προγράμματα μιλάμε, ήταν εκπαίδευση, ήταν κατασκευή αυτοκινητοδρόμων ή ε, άλλες κατασκευές. Δεύτερη ερώτηση, ποια ήταν τα ποσά και κατάφεραν να ανακτηθούν. Τρίτη ερώτηση, λογοδότησε κάποιος και προσήχθη δικαιοσύνη. Και τέταρτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, βάλει εκείνου που ευθύνονται για τι απάτη σε μια μαύρη λίστα για το μέλλον. Αυτές ήταν οι ερωτήσει μου τώρα. Καταγράφεται μια αύξηση στον αριθμό των υποθέσεων ατασταλιών και απάτης που εντοπίστηκαν. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτό οφείλεται σε βελτίωση της διαδικασιών για την ανείχνευση αυτών των υποθέσεων, αλλά κατά την άποψή μου ο αριθμός των εννέα υποθέσεων είναι μάλλον μη ρεαλιστικός. Ο ο ΛΑΦ έχει ξεκινήσει μια, την κατάρτιση μιας νέας μεθοδολογίας για την εντοπισμό της απάτης στον τομέα των δημοσίων ε, ε, ε, προμηθειών και την ποσοτικοποίηση της απάτης. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Μουλτέρ. Μάλτα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η ερώτησή μου δεν έχει τόσο σχέση με τη σημερινή κατάσταση. Πρέπει να συνεχίσουμε τι ε, προσπάθειε μα με κάθε μέσο στη διάθεσή μα για την καταπολέμηση τη απάτηση. Το ερώτημά μου όμω είναι τι μπορούμε να αναμένουμε εάν δημιουργηθεί το γραφείο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Ποια θα είναι η διαφορά, τι θα μπορούσε να κάνει το γραφείο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα που δεν μπορεί να το κάνει ήδη ο Όλαφ. Ή με άλλα λόγια. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα θα, που θα μπορούσαμε να αναμείνουμε από το γραφείο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Πρέπει να πω ότι εγώ πάντα ήμουν υπέρ αυτής της, της δημιουργίας αυτού του γραφείου. Ήμουν και μέλος της Επιτροπής του Κοινοβουλίου ήδη από το 1995 σε Επιτροπή που ε, διερεύνησε υποθέσεις απάτης. Όμως θα ήθελα να μου εξηγήσετε και να μου δώσετε και επιχειρήματα γιατί θα ε, βοηθούσε η δημιουργία ενός γραφείου Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Για να μπορώ και εγώ να υποστηρίξω αυτή την ιδέα ακόμα πιο ένθερμα. Με την άδειά σας ο Πρόεδρος θα ήθελα και εγώ να πω κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα είναι θετικό ότι έχουμε μία συστηματική και τακτική ενημέρωση για αυτές τις ατασταλίες και για την εντοπισμό των απατών. Σας ευχαριστούμε λοιπόν κύριε Σεμέτα που μας δίνετε στοιχεία, αριθμητικά στοιχεία. Δεύτερον, αναφερθήκατε και κάνατε και κάποιες πολιτικές προτάσεις. Πιστεύω και μάλλον είναι προφανές ότι ποτέ δεν θα ολοκληρωθεί ο αγώνας για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς. Είναι στην φύση του ανθρώπου. αλλά χρειάζεται γι' αυτό να έχουμε ισχυρούς μηχανισμούς καταπολέμησης της απάτης και επίσης θα πρέπει και η τιμωρία να είναι παραδειγματική και να λειτουργεί αποτρεπτικά. Και ο τρόπος για να γίνεται αυτό, όπως έκανε η κυρία Μακόη, είναι να αναφερόμαστε ονομαστικά στις χώρες, στα οργανισμούς και στα άτομα που διέπραξαν τέτοιες απάτες, αδικήματα. Κύριε ε, Επίτροπε, θα μας είχατε βοηθήσει και νομίζω όλοι θα ε, ήμασταν ευτυχείς αν είχαμε και γραπτός την ομιλία σας, γιατί είχε και αριθμητικά στοιχεία. Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω τώρα το λόγο για να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ετέθεσαν πριν συνεχίσουμε με τον κύριο Κεσλάρ. Κύριε Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα μετά από τις παρεμβάσεις που έγιναν από τους συναδέλφους να, να θέσω, όπως είπε η κυρία Μακοβέη, το ζήτημα του κόστους της ε, διαφθοράς. Γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο ζητούμε να εξακριβώσουμε. Όταν εξετάζουμε το κόστος του αγώνα κατά της διαφθοράς, είναι χρήσιμο να μπορούμε να ξέρουμε πόσο είναι και το κόστος της διαφθοράς σε μια εποχή που υπάρχουν σημαντικές δημοσιονομικές περικοπές. Επίσης υπάρχει και αυτή η συζήτηση που γίνεται μεταξύ μας. Αν υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ατασταλιών και απατών σε ορισμένα κράτη-μέλη, θεωρείται ότι έχουν ένα πρόβλημα. Αλλά είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις, πάλι κάτι δεν πάει καλά, γιατί δεν ψάχνουν αρκετά τις ε, ατασταλίες ενδεχομένω. Πότε κύριε Επίτροπε, νομίζω <clears throat> μπορείτε να μου πείτε, πότε θα έχουμε την μεθοδολογία που θα μας επιτρέπει, αυτές οι χώρες έχουν κίνδυνο ατασταλιών, αυτές δεν έχουν. Γιατί ή το να έχει κανείς πολλές περιπτώσεις ε, ατασταλιών ή απάτες ή περιπτώσεις αυτού του είδους. Αυτό δεν είναι θετικό, αλλά ούτε είναι θετικό να μην παρουσιάζονται καθόλου τέτοιες περιπτώσεις, γιατί σίγουρα ξέρω ξέρουμε ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, αλλά απλώ δεν εντοπίζονται. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία από πολιτική άποψη είναι ευαίσθητα γιατί δίνουν τροφή στον ευρωσκεπτικισμό και το αντιευρωπαϊκό πνεύμα. Θα ήταν χρήσιμο να έχουμε λοιπόν μια μεθοδολογία που θα μας λέει πράγματι υπάρχει μια δυνατότητα να κρίνουμε πόσο καλή είναι η κατάσταση σε κάθε κράτος μέλος και όταν έχουμε χώρες οι οποίες δεν δίδουν καθόλου δεδομένα να μπορούμε να έχουμε μια δυνατότητα να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις χώρες αυτές. Να μπορέσουμε κάποια στιγμή να εξηγήσουμε στον πολίτη ότι έχουμε ένα σύστημα το οποίο εντοπίζει τα προβλήματα διαφθοράς και ο πολίτης μπορεί να κοιμάται ήσυχο διότι δεν θα υπάρχει διαφθορά στη χώρα του. Και να κάνουμε τη διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών που δίνουν στοιχεία και αυτών που δεν δίνουν στοιχεία. Αλλιώς όλοι θεωρούνται ότι είναι εξίσου κακοί, εξίσου διεφθαρμένοι και επομένως και η κοινή γνώμη θέλει και κάποια θετικά νέα για να μπορέσει να έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας και θέλω να ευχαριστήσω την συγγήτρια για τα θερμά της λόγια σε σχέση με την ετήσια έκθεση της Κομισιόν και με την άποψή σας ότι πράγματι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε την ποιότητα και να παρουσιάσουμε με διάφανο τρόπο τα στοιχεία τα οποία έχουν συγκρίσιμο χαρακτήρα και μας επιτρέπουν να κάνουμε μια σωστή σύγκριση. Μην ξεχάσετε ότι αυτή η έκθεση είναι σε σχέση με τις ατασταλίες και απάτες μάλλον που εντοπίζεται και αναφέρεται από τα κράτη-μέλη. Δηλαδή έχουν ήδη ληφθεί κάποια μέτρα σε σχέση με αυτές τις περιπτώσεις και τα ποσά της, τα κονδύλια που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση είτε έχουν τύχη ανάκτησης ή είναι στο δρόμο της ανάκτησης. Δεν πρέπει λοιπόν να θεωρούμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει αδιαφορία για αυτές τις περιπτώσεις. Επίσης, ε, συμμερίζομαι και εγώ την άποψή σας και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να είμαστε φιλόδοξοι σε ό,τι αφορά την νομοθετική μεταρρύθμιση και με τις δύο αυτές προτάσεις για την εισαγγελική αρχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την οδηγία TIF δημιουργούμε ένα νέο ευρωπαϊκό τοπίο σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτές οι προτάσεις να μην αποδυναμωθούν. Πραγματικά χάρη στην οδηγία TIF η έννοια της ε, απάτης να περιλαμβάνει και το ξέπλυμα χρημάτων και την διαφθορά. Αν γίνουν αυτά δεκτά λοιπόν θα υπάρξει εναρμόνιση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μας δώσει τη δυνατότητα να αποφύγουμε μεγάλες διαφορές στην ερμηνεία διαφόρων ειδών απάτης. Και αυτό λοιπόν θα βοηθήσει πάρα πολύ και τον αγώνα κατά της ε, απάτης. Και για το, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή μας είπε ο κύριος Μίλντερ ποια θα είναι τα κέρδη από μια τέτοια νέα αρχή. Και εγώ ανέφερα ορισμένα από αυτά τα πλεονεκτήματα τα οποία θα προκύψουν σήμερα. Δεν έχουμε καθόλου ένα φορέα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί να αντιμετωπίσει θέματα ποινικού δικαίου. Οπότε καταλήγουμε στην Όλαφ που έχει την αρμοδιότητα για να κάνει διοικητικού χαρακτήρα έρευνες και μετά δίδει τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών στις εθνικές αρχές, συγγνώμη και οι εθνικές αρχές πολλές φορές επαναλαμβάνουν όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει, γιατί στη συνέχεια πρέπει να εφαρμοστεί το εθνικό δίκαιο στην ε, έρευνα αυτή και επομένως οι προσπάθειες που έχουν γίνει από την Όλαφ κατά τη διάρκεια της διοικητικής της έρευνας πολλές φορές πρέπει να επαναληφθούν στα κράτη-μέλη για να μπορέσει να γίνει η δικαστική δίωξη <clears throat> εναντίον αυτών οι οποίοι παρέβησαν το ποινικό δίκαιο. Αυτό χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται χρόνο και δεν είναι πολύ αποτελεσματικό. Με την εισαγγελική αρχή λοιπόν, ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα θα είναι ότι μία έρευνα η οποία θα έχει γίνει από την εισαγγελική αρχή ή τους αναπληρωτές εισαγγελεί στα μελη θα μπορεί να θεωρείται αποδεκτή από όλα τα κρατημέλη ως ένδικη διαδικασία. Ακόμα λοιπόν και αν υπάρχει μία έρευνα που εμπλέκει πέντε κρατημέλη και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έχουν ε, υπάρχουν αποτελέσματα σε σχέση με την έρευνα σε μια χώρα, τη Γερμανία ή τη Γαλλία. Όλα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ω πορίσματα και σε άλλε χώρε όπω είναι η Ιταλία και η Αυστρία και με τον τρόπο αυτό θα έχουμε μια πιο γρήγορη και αποτελεσματική διαδικασία. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή θα πρέπει να έχει όλες τις εξουσίες οι οποίες φυσιολογικά είναι στα χέρια των εθνικών εισαγγελέων και ανακριτών στα κράτη-μέλη. Η οδηγία απαριθμεί τις εξουσίες αυτές που θα πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή, το δικαίωμα ε, ελέγχου και έρευνας σε σπίτια, σε πληροφορικά συστήματα, όλα αυτά τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα σε ποινικέ διαδικασίε και ένα σημαντικό στοιχείο αυτής της πρότασης είναι ότι όλες αυτές οι ενέργειες θα απαιτούν την έγκριση δικαστικών αρχών. Υπάρχει έτσι μια ισορροπία μεταξύ των εξουσιών που έχει ο Ευρωπαίος εισαγγελέα και της ανάγκης προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών που εξασφαλίζεται από τις εθνικές δικαστικές αρχές. Αυτό είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να το τονίσουμε. Ένα τρίτο σημείο. Έχουμε συζητήσει διαμακρών με τα κράτη-μέλη σε σχέση με, με τη σωστή αρχιτεκτονική που θα πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή και αποφασίσαμε ότι δεν θα πρέπει να είμαστε ε, ιδιαίτερα παρεμβατικοί στα εθνικά συστήματα των κρατών μελών. Θα έχουμε λοιπόν το σύστημα αυτό που με ένα Ευρωπαίο εισαγγελέα και θα εκχωρούνται οι εξουσίες τους σε εθνικούς εισαγγελείς οι οποίοι θα εφαρμόσουν και τον εθνικό νόμο της ε, χώρας στην οποία βρίσκονται και ο δικαστικός έλεγχος σε κάθε χώρα θα βασίζεται στην εθνική νομοθεσία. Οπότε και οι δύο πλευρές θα γνωρίζουν την νομοθεσία η οποία ισχύει σε κάθε κράτος μέλος και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να έχουμε μια πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση. Τώρα, αν οι εθνικές αρχές έχουν ερωτήματα σε σχέση με την εφαρμογή του κανονισμού, θα είναι πάντα δυνατό να θέσουν προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε σχέση με την ερμηνεία του Α ή Β κανονισμού. Νομίζω λοιπόν ότι η πρότασή μας εξασφαλίζει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της ανάγκης να αντιμετωπίσουμε σε οριζόντιο επίπεδο την απάτη κατά των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάγκη να είμαστε πιο προσεκτικοί σε σχέση με τον τρόπο που παρεμβαίνουμε στα <clears throat> εθνικά νομικά συστήματα και ίσως όλα αυτά μπορεί να πείσουν τον κύριο Μούλντερ να υποστηρίξει την πρότασή μας σε χρονικό επίπεδο. Σήμερα είναι δύσκολο να προβλέψω πόσος χρόνος θα χρειαστεί, αλλά η Κομισιόν και η Λιθουανική Προεδρία είναι δεσμευμένοι να διοργανώσουν ένα σημαντικό αριθμό συζητήσεων και διαβουλεύσεων κατά τη διάρκεια της Λιθουανικής Προεδρίας για τα θέματα αυτά. Και ξέρετε ότι η συνθήκη προβλέπει μια απλοποιημένη διαδικασία για την ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα αυτό. Πιστεύω λοιπόν ότι τελικά θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ενισχυμένη συνεργασία για τα θέματα αυτά, διότι ξέρουμε ότι κάποια κράτη-μέλη, τουλάχιστον σε αυτό το χρονικό σημείο δεν υποστηρίζουν αυτή την πρόταση. Ίσως όμως κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων θα υποστηρίξουν αυτό το σχέδιο. Η Κομισιόν λοιπόν θέλει να προωθήσει αυτή την πρόταση ώστε να εγκριθεί η απόφαση αυτή το ταχύτερο δυνατό. Κάποια ερωτήματα επίσης για την ε, διαφθορά και τις ε, μνήες που περιέχονται στην έκθεση. Σωστά είπε η κυρία Μακοβέη ότι υπήρχαν 29 9 υποθέσεις διαφθοράς που εντοπίζονται στην έκθεση. Σας λέω όμως και πάλι ότι αυτή η έκθεση βασίζεται στις αναφορές των κρατών μελών αλλά μπορούμε να ζητήσουμε από τα κρατη μας να μας δώσουν πιο πολλές λεπτομέρειες για αυτές τις ε, περιπτώσεις, εφόσον δεν βρίσκονται ακόμα σε, στα πλαίσια συνεχιζόμενης δικαστικής διαδικασίας στα κρατη Και αν δω τώρα το, την ευρύτερη εικόνα για τα θέματα διαφθοράς, την οποία ανέφερε και η κυρία Αγιάλα Σέντερ, εμείς περατώνουμε το, την επεξεργασία μας σε σχέση με την πρώτη έκθεση της Κομισιόν για την διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή η πρόταση θα παρουσιαστεί, η έκθεση μάλλον θα παρουσιαστεί από την Κομισιόν και θα δώσει μια πλήρη εικόνα για την εικόνα της διαφθοράς στα κράτη-μέλη μας και επίσης συστάσεις για τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν ώστε με καλύτερο τρόπο να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό. Η κυρία Μάνστρομ είναι αυτή η οποία είναι η επί της ουσίας αρμόδια για το θέμα αυτό, αλλά και εγώ φυσικά και οι Όλαφ συμβάλλουν σημαντικά σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτό το εγχείρημα και ελπίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα βοηθήσει και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να έχουν μια καλύτερη εικόνα στον τομέα αυτό της διαφθοράς. Και προσβλέπω στη συζήτηση που θα διαμειφθεί σε σχέση με την νέα έκθεση, την πρωτοβουλία της Όλαφ σε σχέση με τη διαφθορά στις δημόσιες προμήθειες και θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό την Τρίτη, την επόμενη Τρίτη, αν θυμάμαι καλά. Θα κάνω και πάλι επίσκεψη στην Επιτροπή σας, δύο φορές αυτή τη βδομάδα, άλλες δύο φορές την επόμενη βδομάδα. Πιστεύω όμως ότι όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα, τα οποία πράγματι πρέπει να μας απασχολήσουν και να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιες λύσεις για όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ αυτά τα οποία είπατε όπως είπα και χτες εμείς χαιρόμαστε να σας έχουμε εδώ πέρα, δεν ξέρω αν χαίρεστε και εσείς να έρχεστε. Αν έχετε χρόνο να ακούσετε και τον κύριο Κέσλερ, κύριε Επίτροπε, μπορεί νομίζω να βρεθεί έτσι, ένα λίγος κοινός τόπος. Μπορώ να μείνω μέχρι τις 11, λέει ο κύριος Επίτροπος. Μέσα μέχρι τις 11 ο κύριος Επίτροπος. Κύριε Γενική Διευθυντά, Τζοβάνι Κέσλερ, του Όλαφ. Τα πράγματα είναι σοβαρά, έχετε το λόγο. Yes, thank you very much. I thank you, Chair and honourable members. Uh, we are. I brought with me a, a, a very, very short and, uh, presentation. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ. Έχω φέρει μια σύντομη παρουσίαση. Και για να δούμε εδώ πέρα. Πρέπει να φανεί στην Maybe, maybe you allow me 30 seconds, uh, Mr. President, while, while the staff of the Parliament is trying to. Λίγη ώρα, αν μπορείτε να μου δώσετε, κύριε Πρόεδρε. Ε, καλά, αν δεν είναι δυνατόν, θα τα πω χωρίς ε, παρουσίαση. Α, μάλιστα, ωραία. Είμαι εδώ πέρα για να σας εξηγήσω το τι κάνει ο Όλαφ ε, σε σχέση με την, ε, να σας παρουσιάσω την έκθεση δραστηριοτήτων του 2012 που βγήκε τον Μάιο και είναι στη διάθεση βεβαίως των μελών. Δεν θα μακρηγορήσω, απλά θα ήθελα να τονίσω κάποια βασικά ζητήματα από τη δραστηριότητα του Όλαφ πέρσι όπως ξέρετε πέρσι ήταν η χρονιά της εφαρμογής ε, μιας εσωτερικής αναδιοργάνωσης που ξεκίνησε από την 1η Φεβρουαρίου του 2012 αναδιοργανώσαμε πλήρως τη Γενική Διεύθυνση. Μάλιστα. Και ξεκινήσαμε κάποιες νέες ερευνητικές ε, διαδικασίες από 1η Φεβρουαρίου. Σας ευχαριστώ. Αυτά θα τονίσω πρώτα. Ήταν λοιπόν μια μεταβατική χρονιά. Και χάρη στην αναδιοργάνωση καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε να κάνουμε κάτι με τις υποθέσεις που χρόνιζαν και είχαν συσσωρευτεί. Το δεύτερο μεγάλο Αντικείμενο της έκθεσης είναι πως ε, το 2012 ήταν η χρονιά στην οποία ο Όλαφ είχε λάβει το μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών, μακράν το μεγαλύτερο αριθμό ε, πληροφοριών ερευνητικού ενδιαφέροντος όπως τις λέμε ε, και τα αιτήματα προήλθαν από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, ε, αρχές των κρατών μελών ε, και ιδιώτες. Κάτι το οποίο δείχνει πόσο χρήσιμος είναι ο Όλαφ και αυτό το θεωρούν και δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς ε, και το κοινό και βεβαίως αυτό είναι μια μεγάλη ευθύνη και βεβαίως και περισσότερη δουλειά. Και το τρίτο βεβαίω είναι η ψηλότερη αποτελεσματικότητα. Καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε, όπως σας είπα, αυτό το πολύ μεγάλο αριθμό υποθέσεων και βεβαίως να ξεκαθαρίσουμε τις υποθέσεις που χρόνιζαν και να τις μειώσουμε κατά πολύ, αλλά να μειώσουμε και τη μέση διάρκεια α, διεκπαιρέωσης μιας υπόθεσης. Εδώ πέρα έχετε τον αριθμό, τους αριθμούς της δραστηριότητάς μας. Βλέπετε στη βάση της πυραμίδας τις πληροφορίες που είχαμε. 2011 ήταν το προηγούμενο ρεκόρ Όλα δεν είχε λάβει τόσες πολλές ε, πληροφορίες μέχρι τότε, 1046. Το 2012 λάβαμε σχεδόν 20% παραπάνω ε, τέτοιες πληροφορίες. Αυτό σημαίνει βεβαίως 20% περισσότερες υποθέσεις που άνοιξαν. Αντιλαμβάνεστε πως το 2012 κλείσαμε 465 έρευνες, όπως λέγεται, πάνω από τις διπλές δηλαδή σε σχέση με τις πλάσεις, σε σχέση με το 2011 και βλέπετε πως παρόλα αυτά φτάσαμε και ε, τις 200 σχεδόν συστάσεις προς τα κράτη-μέλη, τα θεσμικά όργανα κτλ. Να τονίσω επίσης κάτι για την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας. Καταφέραμε να μειώσουμε τη διάρκεια της φάσης επιλογής, την πρώτη φάση δηλαδή επεξεργασίας της ερχόμενης πληροφορίας και τη φάση στην οποία λαμβάνεται η απόφαση για το αν θα ξεκινήσει ή όχι μια έρευνα. Πάρα πολύ σημαντική φάση και πρέπει να είναι σύντομη γιατί οι εταίροι μας, ειδικά οι αρχές των κρατών μελών ή τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να γνωρίζουν και σύντομα το εάν θα ξεκινήσει μια έρευνα ο Όλαφ ή όχι για οποιονδήποτε λόγο. Από όταν λοιπόν 1η Φεβρουαρίου πέρσι συστάθηκε μια ειδική ομάδα καταφέραμε να μειώσουμε δραματικά τη διάρκεια αυτής της ε, πρώτης φάσης σε 1,5 μήνα. Και μπορώ να σας πω πως ε, αυτή η μέση διάρκεια ισχύει και για το 2013. Οπότε Όλαφ μπορεί να δώσει μια απάντηση στις αρχές για το εάν θα ξεκινήσει ή όχι μια έρευνα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και αυτό βέβαια το εκτιμούν ιδιαίτερα οι εταίροι μας. Βλέπετε επίσης στη διαφάνεια αυτή, ε, όλες αυτές οι διαφάνειες είναι από την έκθεση επί τη ευκαιρία που έχετε. Βλέπετε εδώ πώς καταφέραμε να αντιστρέψουμε την αυξητική τάση που υπήρχε όσον αφορά τη διάρκεια της έρευνας και το 2012 ακόμα και αν είχαμε υψηλότερο αριθμό ερευνών καταφέραμε να μειώσουμε σοβαρά τη συνολική διάρκεια των ε, υποθέσεων. Και επίσης μπορώ να προβλέψω πως αυτή η τάση θα συνεχιστεί και το 2013. Αυτές είναι λοιπόν οι έρευνες ε, που συνεχίζονται μέχρι το τέλος του έτους για να αποκτήσετε μια ιδέα. Βλέπετε πως οι περισσότερες από αυτές αφορούν τα διαρθρωτικά ταμεία. Επίσης την εξωτερική βοήθεια και αρκετά σημαντικό αριθμό 90 υποθέσεις αφορούσαν τις λεγόμενες εσωτερικές έρευνες, ε, προσωπικό δηλαδή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα θα ήθελα να δώσω κάποιες πληροφορίες που και ε, αυτό αφορά τις πληροφορίες που λαμβάνουμε. Υπάρχει νομίζω λοιπόν αύξηση των πληροφοριών που λαμβάνει όλα. Το 2012 ήταν ε, έτος ρεκόρ και τώρα αναλύσαμε συνοπτικά την πηγή των πληροφοριών. Όπως βλέπετε, κατά τη διάρκεια των ετών, βλέπετε την κίτρινη γραμμή οι πληροφορίες από ιδιώτες αυξάνονται. Φτάσαμε τις 889. Κάτι εδώ πέρα τα λέω από ιδιώτες ε, συμπεριλαμβάνει και τις ανώνυμες πηγές. Ε, αλλά σημαντικότερη επίσης είναι η μπλε γραμμή βλέπετε πως πέρσι καταφέραμε να αντιστρέψουμε μία ανησυχητική τάση που ήταν η μείωση επί σειρά ετών των πληροφοριών από τις δημόσιες αρχές, δηλαδή ε, αστυνομία και δικαστήρια κρατών μελών, οι ελεγκτικές αρχές κρατών μελών και τα θεσμικά όργανα. Βλέπετε πως μετά από πολλά χρόνια είχαμε σημαντική αύξηση των ε, καταγγελιών, των πληροφοριών από τα κρατη Κάτι το οποίο μας δείχνει μία διάθεση για συνεργασία από τις ε, αρχές και επίσης την εμπιστοσύνη σαν Όλαφ. Εάν ζητήσει κανείς πληροφορίες στον Όλαφ, ε, εάν στείλει κανείς πληροφορίες στον Όλαφ, σημαίνει πως υπάρχει εμπιστοσύνη στον Όλαφ. Βλέπετε εδώ πέρα πως σε τι αντιστοιχεί η μπλε Ε, δηλαδή βλέπετε την ανάλυση μεταξύ ε, αρχών κρατών μελών και ε, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Και βλέπετε πως η αύξηση ε, οφείλεται στις εθνικές αρχές. Και βεβαίως στα θεσμικά όργανα. Τέλος. Για πρώτη φορά βλέπετε εδώ πέρα πιο λεπτομερός, το βλέπετε και στη γραπτή έκθεση. Προσπαθήσαμε να δούμε τις πληροφορίες από τα κράτη-μέλη. Εδώ πέρα βεβαίως δεν έχετε τις ε, ανώνυμες ε, πηγές. Ε, βεβαίως οι ανώνυμες, οι ανώνυμες πηγές δεν πάνε σε κάποιο κράτος μέλος, ούτε και κάποιοι που κάνουν ε, καταγγελία εσωτερική. Αλλά ενδιαφέρον είναι να δούμε πως οι δύο χώρες, η Γερμανία και η Ιταλία, είναι σχεδόν το μισό των πληροφοριών που λαμβάνουμε από τις δημόσιες ε, αρχές. Θεωρούμε πως όσο, όσα περισσότερα αναφέρουν ε, τα κράτη-μέλη, κάτι τέτοιο σημαίνει πως ε, τόσο και μεγαλύτερη αντίδραση υπάρχει στην απάτη. Ειδικά δηλαδή οι γερμανικές αρχές ε, συνεργάζονται μαζί μας ε, ε, συνεχώς στην καταπολέμηση της απάτης. Ενδιαφέρον είναι να συγκρίνουμε πώς πληροφορίες λαμβάνουμε σε ένα κράτος μέλος από τις δημόσιες αρχές σε σχέση με το τι λαμβάνουμε από τον ιδιωτικό τομέα. Ε, τώρα την ερμηνεία θα την κάνετε εσείς, αλλά είναι σημαντικά νομίζω τα δεδομένα, γιατί αν ένα κράτος μέλος π.χ. δεν λαμβάνουμε πληροφορίες από τις δημόσιες αρχές και έχουμε πολλές ε, καταγγελίες ε, από ιδιώτες, όπου είναι έτσι μπορεί να είναι επιχειρηματίες. Οποιοςδήποτε ιδιώτης, η κοινωνία των πολιτών να καταγγέλει πιθανή απάτη, σημαίνει πως ίσως υπάρχει πρόβλημα. Ε, είναι πολύ ενδιαφέροντα νομίζω αυτά τα δεδομένα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και για τον Όλαφ. Είναι χρήσιμα για μας για να δούμε που πρέπει να ρίξουμε περισσότερο βάρος για να έχουμε καλύτερη συνεργασία. ανταυτού θα έλεγα ε, πως αυτό είναι πιο χρήσιμο για εμάς και για εσάς νομίζω αντί να έχουμε τον συνήθι πίνακα των κρατών μελών με τον αριθμό των ερευνών σε κάθε χώρα. Ε, επί τη ευκαιρία, πρώτα απ' όλα είναι πολύ δύσκολο ε, να ε, κάνουμε αυτή την κατανομή ανά κράτος μέλος, γιατί Κάποιες έρευνες περιορίζονται σε ένα κράτος μέλος, αλλά οι περισσότερες είναι δύσκολο να εντοπιστούν σε μία χώρα μόνο. Κατά κανόνα δηλαδή, ε, μία έρευνα απαιτεί δραστηριότητα σε πολλά κράτη-μέλη. Και κάποιες από τις έρευνές μας είναι, θα έλεγα, εκφύσεως ευρωπαϊκές και είναι δύσκολο να ε, εντοπιστούν σε ένα κράτος μέλος. Και στο παρελθόν είχαμε κάποιες παρεξηγήσεις ε, όσον αφορά την ερμηνεία αυτών των στοιχείων. Παραδείγματος χάρη το Βέλγιο ήταν πάντα η χώρα που ερευνούσαν περισσότερο. Αλλά τι έγινε, βάζαμε το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Βέλγιο. Αυτό δεν λέει τίποτα για τους Βέλγους βεβαίως και το, το Βέλγιο ως χώρα. Έτσι. Και διάφορα τέτοια πράγματα, πιθανές παρερμηνίες. Ακριβώ γιατί δεν υπήρχε η σωστή ερμηνεία των δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικά για τον Όλαφ, ε, όχι μόνο για τον Όλαφ, αλλά και για να δούμε και τη δυνατότητα των κρατών μελών ε, να αντιδράσουμε. Θα λοιπόν να τελειώσω εδώ πέρα και να σας διαβεβαιώσω πως ε, καταφέραμε το 2012 ε, να επιφέρουμε μεγάλες αλλαγές στις διαδικασίες του Όλαφ με νέες ερευνητικές διαδικασίες για να ευθυγραμμιστούμε ήδη με αυτά τα οποία θα προβλέπει ο νέος κανονισμός. Καταφέραμε να διάσουμε τα συρτάρια και τις υποθέσεις που είχαν συσσωρευτεί. Το προσωπικό μας ε, Ε, όλο το προσωπικό, όχι μόνο το ερευνητικό προσωπικό, είχε πραγματικά τεράστιο φόρτο εργασίας, τεράστιο αριθμό υποθέσεων που κατάφερε να κλείσει και να καταφέρει να αντιδρά η υπηρεσία μας ε, πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Και αυτά ισχύουν και για το 2013, θα τα ξαναπούμε σε λίγους μήνες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Γενική Διευθυντά. Τώρα περνάμε στη συζήτηση. Κυρία Γκρέσλε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη που δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω όλη την παρουσίαση, αλλά έπρεπε να είμαι σε μια άλλη επιτροπή. από τα στοιχεία αυτά του 2012 νομίζω ότι έχουμε ορισμένα στοιχεία τα οποία μας ενδιαφέρουν. Το 2012 όμως ήταν μια χρονιά που έγιναν πολλά, ε, υπάρχουν κάποιες στατιστικές ανομαλίες ούτως είπε γιατί υπήρξαν πολλές μεταφορές οι οποίες έλαβαν χώρα Υπήρξαν 21 περιπτώσεις οι οποίες έχουν κλείσει και θα ήθελα να ξέρω σε αυτές τις περιπτώσεις αν ξανά άνοιξαν αυτές οι έρευνες. Και δεν ξέρω πώς έγινε δυνατόν να κλείσαν όλες αυτές τις περιπτώσεις μέσα σε μία μέρα οι υποθέσεις και να ξανά ανοίξουν πάλι σε μια μέρα. Υπάρχουν κάποιες νομικές προϋποθέσεις για να ξεκινήσει και πάλι μια υπόθεση και δεν βλέπω πόσο εύκολο είναι να έχει γίνει κάτι τέτοιο για ένα τόσο μεγάλο αριθμό ε, υποθέσεων επίσης. Κάτι το οποίο είχε μεγάλη σημασία για πολλά χρόνια για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα της Όλαφ είναι να αντιμετωπίσουμε την συνέχεια που δόθηκε. Ποιες περιπτώσεις λοιπόν έχουν κλείσει αλλά υπήρξε μια συνέχεια είτε δι... διοικητικές συνέπειες είτε πειθαρχικές ε, ε, διαδικασίες είτε ποινικέ διαδικασίες. Πόσες είναι οι περιπτώσεις λοιπόν που είχαν κάποιο αποτέλεσμα. Είχαμε λοιπόν τέτοιες υποθέσεις το, τον ίδιο αριθμό το 2012 όπως και το 2011. 100 περιπτώσεις που δόθηκε συνέχεια σε αυτές. Δεν μπορώ λοιπόν να κατανοήσω πού βρίσκεται η επιτυχία τη ΣΟΛΑΦ έναντι του 2011 όταν δεν μπορώ να ανοιχνεύσω στα, στους αριθμούς αυτήν την επιτυχία σε ό,τι αφορά πράγματος χάρη. Και υπάρχουν και κάποια στρεβλωτικά στοιχεία τα οποία αλλάζουν τους αριθμούς λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του 2012. Ίσως θα πρέπει να υπάρξει και μια αλλαγή στην ονοματολογία που χρησιμοποιείται για να είναι πιο σαφή τα πράγματα, γιατί η Κομισιόν πολλές φορές χρησιμοποιεί Ε, και οδηγεί στο να μπορεί η Όλαφ να κάνει δηλώσει τις οποίες δεν μπορεί να τεκμηριώσει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να πω λοιπόν, εγώ προσπάθησα να ελέγξω και πάλι τα στατιστικά στοιχεία, αλλά αυτό το οποίο διαπιστώνει κανείς είναι ότι είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές αυτές οι στατιστικές για το πόσες συνεντεύξεις έγιναν με τους εμπλεκόμενους επιτόπιες έρευνες, έρευνες με υπολογιστή. Σε μία από τις 20 περιπτώσεις έχετε κάνει μονάχα σε μία από τις 20 περιπτώσεις δεν ακούσατε τον ε, ενδιαφερόμενο. Και δεν θέλω τώρα να αναφερθώ για την περίπτωση Ντάλι, του Επιτρόπου κ. Ντάλι. 7,5% όλων των ε, συνεντεύξεων που έκανε η Όλαφ ήταν με εμπλεκόμενη στην υπόθεση Ντάλι, 9% για ελέγχους στα γραφεία, των ελέγχων έγινε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίπτωση αυτή. Λοιπόν, αν βασιστούμε σε αυτό, τι μένει για, το, για τις υπόλοιπε έρευνες της Όλαφ και πώς εξασφαλίζεται τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι γίνεται με όλες αυτές τις υποθέσεις οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο της Όλαφ και εμπίπτουν στην ε, παραγραφή. Και τι έγινε με όλες αυτές τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν έχει αναλυθεί καμία ενέργεια. Θα ήθελα λοιπόν να ξαναδούμε τη μονάδα όμικρον 1 όπου υπήρξε μια αναδιοργάνωση. Θα ήθελα να ξέρω πόσο αποτελεσματική είναι η λειτουργία αυτής της μονάδος και θα ήταν χρήσιμο να μας δώσετε και κάποια στοιχεία για όλα αυτά. Ευχαριστώ. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ. Αρκετά ερωτήματα θέσατε. Και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Σόντεργαρτ. Σας ευχαριστούμε για την έκθεση. Θα ήθελα κάποιες επιπλέον πληροφορίες, κύριε Κέσλερ, για το ποια είναι η διαφορά μεταξύ των πληροφοριών που σας έρχονται από τις ε, κρατικές αρχές αφενός και τις ε, πληροφορίες που σας έρχονται από, από τους ιδιώτες. Λοιπόν, έλεγα, υπήρξε κάποιο μικρό πρόβλημα με τη διερμηνία. Επαναλαμβάνει ο μιλητή. Σα ευχαριστώ για τι ε, πληροφορίε που μα δώσατε. Απλώ θα ήθελα να εμβαθύνουμε λίγο. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε περισσότερο και καλύτερα ποια είναι η διαφορά μεταξύ των πληροφοριών που λαμβάνετε από τι κρατικέ αρχέ και από του ιδιώτε. γιατί πρέπει να πω ότι είμαι έκπληκτος ε, κοιτώντας αυτά τα στοιχεία. Και γιατί αυτό, γιατί διαπιστώνω ότι από ορισμένα κράτη-μέλη δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από τις κρατικές αρχές, ενώ από ιδιώτες υποβάλλονται σχεδόν διπλές-τριπλές καταγγελίες σε αριθμό. Θα ήθελα κάπως να ε, μου εξηγήσετε γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί σε ορισμένε περιπτώσει είναι οι ιδιώτε που, παρέχουν περισσότερε πληροφορίε στον Όλαφ. Ένα παράδειγμα είναι η Ουγγαρία. Στην Ουγγαρία είχαμε μία περίπτωση, μία υπόθεση από τι κρατικέ αρχέ και 17 καταγγελίες από ιδιώτε. Δεν είναι εκπληκτική αυτή η διαφορά. Θα ήθελα να μου την εξηγήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στην εισηγητριά, την κυρία Αγιάλα Σάντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον κύριο Κέσλερ για τις πληροφορίες που μας έχει δώσει και τις ε, προσπάθειες που έχει καταβάλει η όλα σε σχέση με τις αιτήσει της Επιτροπής μας στις προηγούμενες ε, συζητήσεις που είχαμε για την ανάγκη να βελτιωθεί και η λειτουργία της ΟΛΑΦ <clears throat> σε όλους τους τομείς και φυσικά σε ό,τι αφορά και τα, τα στοιχεία, τα δικαιώματα των υποκείμενων σε έρευνες κτλ. Έχουμε λοιπόν ένα, μια διαφορετική εικόνα την οποία έχουμε πια σε σχέση με τους κινδύνους μετά από αυτά τα οποία μας έχει πει η Όλαφ και έχουμε και νέους, νέες εικόνες σε σχέση με τη λειτουργία της υπηρεσίας σας. Είπατε προηγουμένως ότι από το 2011 μέχρι το 2012 έλαβε χώρα μια αναδιοργάνωση σε εσωτερικό επίπεδο, ήταν ένα μεταβατικό έτος και αναφερθήκατε και στο ξεκαθάρισμα υποθέσεων. Θα ήθελα να καταλάβω λοιπόν πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία. Είπατε ότι έχουν αυξηθεί επίσης οι πληροφορίες που λάβατε, γιατί είναι θετικό αυτό, γιατί αυτό δείχνει ότι γίνεται πιο γνωστή η Όλαφ και είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να βελτιώσει τον έλεγχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω μεταξύ των περιπτώσεων που είναι ανοιχτέ και αυτών που είναι υπό επεξεργασία το 2011, εγώ δεν ξέρω καλά μαθηματικά διότι με τον Ανθρωπιστικό σπουδών, είπατε ότι είναι περίπου 200 περιπτώσεις και το διπλό έχουμε το 2012 σε ανοιχτέ περιπτώσεις και περιπτώσεις οι οποίες είναι υπό έρευνα. Τι σημαίνει αυτό. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ανοιχτές και υποεξέταση εξέταση περιπτώσεις. Επομένως, η εκαθάριση των υποθέσεων που λέτε είναι περισσότερο ένα θέμα οργάνωσης. Η επιλογή που γίνεται των υποθέσεων που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει γίνει καλά η επιλογή αυτών των υποθέσεων. Έχουν μειωθεί οι <clears throat> σε σχέση με το αν θα επιλεγεί ή όχι μια περίπτωση, αλλά το, το όγκος εργασίας φαίνεται ότι παραμένει, δεν έχει αλλάξει. Στις περιπτώσεις αυτές λοιπόν βλέπω αυτή τη μεγάλη διαφορά και ποια είναι η διάρκεια εξέτασης μέχρι να κλείσει μια υπόθεση. Επίσης, σε σχέση με την λειτουργικότητα του προσωπικού της ΟΛΑΒ, ξέρω ότι έχετε κάνει μια προσπάθεια να μπορέσετε να προσλάβετε προσωπικό το οποίο θα εστιάσει περισσότερο το έργο του στις έρευνες που ενδιαφέρουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά τι σημαίνει αυτό η αρρωγή προς τις έρευνες οι οποίες ε, είναι εν εξελίξει, δεν έχω καταλάβει ακόμα. <clears throat> και λέτε επίσης ότι υπάρχει και εξωτερικό προσωπικό το οποίο ασχολείται με τις έρευνες. Τι είναι, είναι εθνικοί εμπειρογνώμονες ή είναι άλλου είδους προσωπικό το οποίο εργάζεται σε αυτές τις έρευνες. Μας κάνετε και μια καλή ε, παρουσίαση για τις νέες δυνατότητες για την ε, βελτίωση του έργου της ΟΛΑΦ και μας λέτε ότι έχετε πάρει πληροφορίες από διάφορα κράτη-μέλη, αλλά θα θέλαμε να ξέρουμε από πού προέρχονται αυτές οι, αυτές οι πληροφορίες. Σίγουρα από την δική μου χώρα θα υπήρχαν πολλές καταγγελίες, αλλά στις πληροφορίες που μας δίνετε δεν αναφέρετε τους καταγγέλλοντες, τους whistleblowers και αυτές που είναι ανώνυμες καταγγελίες. Θα θέλαμε όμως να ξέρουμε τι γίνεται για αυτές τις περιπτώσεις, αν προέρχονται από τις κρατικές υπηρεσίες ή από καταγγέλλοντες whistleblowers. Θα μας έδινε μια πολύ καλύτερη ιδέα. Επίσης, όπως είπε ο κύριος ε, Σόντεργατ, είναι απαραίτητο να υπάρχει και πάλι εμπιστοσύνη μεταξύ των διοικητικών αρχών ότι γίνεται σωστά το έργο της. Όλα αυτά ήθελα να σας ρωτήσω αν με τη συνεργασία σας στις χώρες, με τις χώρες αυτές όπου δεν υπάρχει καμία καταγγελία από τις δημόσιες αρχές, αν σημαίνει αυτό ότι λειτουργεί καλά η συνεργασία ή ότι υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα. Και επίσης θα ήθελα να ξέρω γιατί δεν υπάρχουν πληροφορίες, ίσως εγώ δεν καταφέρω να τη δω. Ποιες υποθέσεις είναι αυτή τη στιγμή τώρα ανοιχτές στα, στα δικαστήρια και πώς προσλαμβάνει προσωπικό η ΟΛΑΦ. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και για την εμπιστοσύνη των πολιτών μας να τους δώσουμε αυτές τις πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια. Είχαμε πολλά ερωτήματα και πολλούς ομιλητές. Ε, κύριε Σεμέτα, πρέπει να ε, μας εγκαταλείψετε. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Και δίνω το λόγο στον ε, Γενικό Διευθυντή του Όλοφ για να απαντήσει. Κύριο Κέσλερ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ ειλικρινά, γιατί όλες αυτές οι ερωτήσεις, όλες αυτές οι παρατηρήσεις μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τι περιμένετε από εμάς. Και τι πρέπει να κάνουμε όσο μπορούμε. Κάποιες διευκρινήσεις σε σχέση με τους αριθμούς. Θα με βοηθούσε αν μπορούσαμε να ξαναέχουμε ε, μια διαφάνεια στις οθόνες. Θα αρχίσω να απαντώ στις ε, ερωτήσεις. Οι πυραμίδες, η διαφάνεια με τις πυραμίδες που σας ε, έδειξα, δείχνουν την χρονική εξέλιξη της ερεύνησης των υποθέσεων. Περίπου 400 υποθέσεις έκλεισαν και άνοιξαν την ίδια μέρα. Πώ το πρωί. Με μια απόφαση του, διευθυντή της Όλαφ, όπω προβλέπεται στον κανονισμό τη Όλαφ. Πρώτα απ' όλα να πω ότι τα στατιστικά στοιχεία έχουν συνταχθεί με τρόπο διαφανή και είναι ορθά. Δεν θα ήθελα να τα αμφισβητήσουμε αυτά, δεν θα ήταν σωστό απέναντι στους έντιμους ε, υπαλλήλους της Όλαφ που τα συνέλεξαν. Στην σελίδα 18 της έντυπης έκθεσης του Όλαφ διευκρινίζεται με σαφήνεια ότι 419 υποθέσεις άνοιξαν ως αποτέλεσμα της αναδιοργάνωσης. αυτός ο μεγάλος αριθμός 718 ε, ε, υποθέσεις που βρίσκονται στο στάδιο του συντονισμού είναι, προέρχεται από εκείνες που ήταν ήδη ανοιχτές συν τις 419 που άνοιξαν 1η Φεβρουαρίου εκείνη την ημέρα άρχισε να ισχύει το νέο οργανόγραμμα και οι νέες διαδικασίες. Αυτές οι 419 υποθέσεις λοιπόν είναι το αποτέλεσμα της μεγάλης προσπάθειας που έγινε καθ' όλη τη διάρκεια του 2011 από την ε, μονάδα που ήταν υπεύθυνη για την ε, επιλογή των υποθέσεων η οποία ανέτρεξε στις υποθέσεις που χρόνιζαν. Κυρίως εκείνες. Ήταν δύσκολο να βρούμε μια ισορροπία γιατί έπρεπε φαινός να ασχοληθούμε με όλες αυτές τις ε, υποθέσεις που χρόνιζαν. Δεχόμασταν κριτική για το γεγονό ότι υπήρχαν τόσες πολλές υποθέσεις που χρόνιζαν. Αλλά ταυτόχρονα, φετερού, έπρεπε να μην ε, σταματήσουμε να ασχολούμαστε με τις νέες υποθέσεις γιατί θα άρχιζαν εκείνες πλέον να συσσωρεύονται, καινούριε. Το αντιμετωπίσαμε αυτό χωρίζοντα το προσωπικό στα κάποιοι ασχολιόντουσαν με τις παλιές υποθέσεις και κάποιοι με τις καινούργιες. Οι 419 λοιπόν υποθέσεις οι οποίες άνοιξαν 1η Φεβρουαρίου, είναι εκείνε που επέλεξε η φεβρουαριου ειναι εκεινες επιλογή μοναδα επιλογης υποθεσεων και θεωρήθηκε σωστό, επειδή υπήρχαν οι ε, νομικές προϋποθέσεις, να ξεκινήσει μια διαδικασία έρευνας ή συντονισμού. Δεν το κάναμε αυτό για να έχουμε ομορφότερα στατιστικά στοιχεία. Εξάλλου δεν κρίνεται το έργο της Όλαφ από τον αριθμό των υποθέσεων που ανοίγει. Κατά την άποψή μου αυτό που μετράει είναι πόσες υποθέσεις καταφέρνει η υπηρεσία να κλείνει με τον σωστό τρόπο και μετά από μια ορθή διερεύνηση. Αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Και είναι κάτι που συμβαίνει μόνο μια φορά. Μόνο μια φορά θα, συμβεί αυτή η αναδιοργάνωση. Φέτος, το 2013, μπορώ ήδη να σας πω ότι μειώνεται ο χρόνος που χρειάζεται για ε, μια ε, διαρεύνηση. Η κυρία Κρέσλε αναφερθήκατε σε κάποιες υποθέσεις follow-up στις οποίες γίνεται, δίνεται συνέχεια σε μια διερεύνηση μπορεί να αποδειχθεί η αθότητα κάποιου κατηγορούμενου. Αυτό δεν το θεωρεί αποτυχία Όλαφ. Θα έλεγα ότι μάλλον θα έπρεπε να ανησυχούμε εάν οι υποθέσεις τις οποίες αποδεικνύεται αθότητα τις θεωρούσαμε αποτυχία. Ή εάν διαπιστωθεί ότι δεν διαπράχθη απάτη. Άρα για εμάς, για τον Όλαφ, η επιτυχημένη έρευνα είναι εκείνη η οποία κατάφερε να διαπισκριβώσει την πραγματικότητα, την αλήθεια. Μπορούμε επίσης να κοιτάξουμε τον αριθμό των συστάσεων που απευθύνουμε προς διοικητικές κρατικές αρχές. Μπορεί να είναι ε, συστάσεις οι οποίες ζητούν δημοσιονομική διόρθωση ή μπορεί επίσης να είναι μιας ε, πληροφορίες προς τις διοκτικές αρχές τις οποίες υποβάλλουμε προς τις δικαστικές διοκτικές αρχές για να εξετάσουν εκείνε αν θέλουν να προχωρήσουν με μια ποινική δίωξη. Πέρσι λοιπόν, όπως σας είπα, ασχοληθήκαμε κυρίως με τις παλιές υποθέσεις, υποθέσεις που χρόνιζαν. Τέσσερα, πέντε χρόνια ή και περισσότερο. Παλιές υποθέσεις. Είναι λοιπόν λογικό ότι όταν ασχολείται με παλιές υποθέσεις δεν θα έχει ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Ίσως αυτό να οδήγησε στη μείωση του αριθμού των συστάσεων. Αν και αν κοιτάξετε την κορυφή της πυραμίδας, το 2012 κάναμε 199 συστάσεις σε σχέση με 175 το 2011. Άρα, ακόμα και ασχολούμενοι με τις παλαιότερες υποθέσεις, τα φέραμε να εντοπίσουμε τα θέματα που κατά την άποψη του Όλεφ θα έπρεπε να ε, ε, τύχουν ε, ενεργειών σε διοικητικό, οικονομικό ή και δικαστικό επίπεδο. Και μπορώ να συνημερώσω ενημερώσω και να προβλέψω ότι το αριθμός των συστάσεων θα είναι ακόμα μεγαλύτερο το 2013. Μπορώ επίσης να προσθέσω, ακόμα και αν δεν το έθιξαν αυτό τα μέλη του Κοινοβουλίου, ότι η Όλαφ επιδιώκει να βελτιώσει το υποπτίας και παρακολούθησης των ενεργειών που αναλαμβάνουν οι διοικητικέ αρχές, οι αρχές οικονομικής διαχείρισης, οι δικαστικές αρχές μετά από τις συστάσεις του Όλαφ. Προσπαθούμε δηλαδή να παρακολουθήσουμε τι συμβαίνει μετά από μια σύσταση δική μας. Αυτό είναι εξάλλου υποχρέωση του Όλαφ ε, με βάση την εντολή, τη νέα εντολή που προβλέπεται για αυτόν ε, στην, ε, στη νέα οδηγία που θα ισχύσει. Ε, τις επόμενες ημέρες. Οφείλουμε να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε τη μη συμμόρφωση. Γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει να παρακολουθούμε και να καταγράφουμε εάν υπάρχει συμμόρφωση ή αν δεν υπάρχει συμμόρφωση από τις αρχές των κρατών μελών στις, συστάσεις μας, στον αυξανόμενο αριθμό συστάσεων που τους απευθύνουμε δεν μπορούμε να τους αναγκάσουμε να αναλάβουν δράση, αλλά τουλάχιστον παρακολουθούμε εάν το πράττουν. Στο νέο κανονισμό υπάρχει ένα στοιχείο που θα μας δώσει τη δυνατότητα ε, να τους ζητούμε αυτά τα στοιχεία, αλλά στον παλαιότερο κανονισμό ε, πρέπει να πούμε ότι δεν είχαμε τέτοιες αρμοδιότητες, δεν είχαμε τη δυνατότητα να απαιτήσουμε στοιχεία, επομένως κάναμε ό,τι μπορούσαμε για την παρακολούθηση. Και είναι δύσκολο να, είχα, να συλλέξει κανείς συστηματικά στοιχεία με αυτόν τον τρόπο. Του χρόνου θα έχουμε τη δυνατότητα να σας ενημερώσουμε καλύτερα όσον αφορά την υλοποίηση, την εφαρμογή των συστάσεων του Όλαφ, κάτι που φαντάζομαι θα βοηθήσει και εσάς στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Αναφερθήκατε στις ανακρίσεις και στις υποθέσεις ε, Ντάλι. Η υπόθεση Ντάλι ήταν μία από τις εκατοντάδε υποθέσεις με τις οποίες ασχολήθηκε ο Όλαφ πέρυσι. Δεν κατάλαβα ακριβώ τι θέλατε να πείτε. Κυρία Γκρέσλε, μας προσάπτεται ότι διεξήγαμε πολλές ανακρίσεις, πολλές συνεντεύξεις με εμπλεκόμενους στην υπόθεση Ντάλι, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε τους δώσαμε τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους, να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, ίσως το παρακάναμε. Αλλά όλες μας οι ενέργειες έγιναν με γνώμονα την ε, προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων αυτών των προσώπων. Ε, ίσως αυτό που μας προσάπτεται είναι ότι κάναμε πολλά για το θέμα του Ντάλι και όχι αρκετά στις υπόλοιπες υποθέσεις. εν πάση περιπτώσει γνωρίζετε ότι δεν είχαμε υποχρέωση να ε, ε, ενεργήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτές οι νέες υποχρεώσεις ε, προβλέπονται τον νέο κανονισμό που θα αρχίσει να ισχύει από 1η Οκτωβρίου 2013. Αλλά πάντως σε κάθε περίπτωση δίνουμε την δυνατότητα στους εμπλεκόμενους να εκφράσουν την θέση τους και να υποστηρίξουν την άποψή τους, να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Είτε μέσω μιας συνέντευξης, όπως συνέβη και δεν το μετανιώνω στην υπόθεση του ε, Τάλι, είτε αποστέλλοντας ε, γραπτός στον εμπλεκόμενο, στον ενδιαφερόμενο, ε, την περιγραφή της υπόθεσης και ζητώντας του να υποβάλει γραπτός ένα υπόμνημα. Ίσως του χρόνου θα ήταν σκόπιμο να συμπεριλάβουμε στα στατιστικά μας στοιχεία ε, πληροφορίες για αυτή τη διαδικασία. Πόσες φορές ζητήθηκε γραπτή ενημέρωση από κάποιον και πόσες φορές ε, τα πρόσωπα αυτά απάντησαν γραπτός. Στο νέο κανονισμό υπάρχουν πλέον πρόνοιες έτσι ώστε όχι μόνο στην υπόθεση Ντάλε αλλά σε όλες τις υποθέσεις να δίνεται δυνατότητα ε, στους εμπλεκόμενους να συνομιλούν με τον Όλαφ, να υποστηρίζουν τις θέσεις τους και να υπερασπίζονται τον εαυτό τους. Πάντα βοηθά τους ερευνητές του Όλαφ να έχουν ε, στη διάθεσή τους και τη θέση ε, των προσώπων αυτών. Με ρωτάτε πώς μπορούμε να μετρήσουμε την επιτυχία. Θα σας δώσω έναν αριθμό που βρίσκεται στην ετήσια, στην ετήσια έκθεση τη γραπτή και αυτός ο αριθμός είναι η μέση διάρκεια που χρειάζεται για την επιλογή μιας υπόθεσης. Δηλαδή πόσο χρόνο χρειάζεται όλα για να αποφασίσει αν μια υπόθεση χρήζει διερεύνηση ή όχι. Καταφέραμε να μειώσουμε αυτή τη διάρκεια από 6, είχε φτάσει 6,8 μήνες πρόπερση σε 1,5 μήνα. Το 2013 αναμένω ότι αυτός ο ρυθμός θα, γίνει, θα φτάσει το 1,6 αλλά σε κάθε περίπτωση ο στόχος μας είναι η, διάρκεια αυτή, η μέση διάρκεια αυτή να παραμείνει μικρότερη από δύο μήνες. Και ο τρόπος που το πετύχαμε αυτό ήταν η δημιουργία μιας ειδική μονάδας επιφορτισμένης με την επιλογή των υποθέσεων, η οποία απαντά γρήγορα, όσο πιο γρήγορα μπορεί, στον, στις αρχές, στον καταγγέλλοντα, εάν όλα αυτά αναλάβει τη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης. Αυτό επίσης ελάφρυνε και το φόρτο εργασία των ερευνητικών ομάδων. Γιατί πριν τη δημιουργία αυτής της ειδική μονάδας, οι ίδιες οι ερευνητικές ομάδες έπρεπε όχι μόνο να διερευνούν έρευνες, αλλά ταυτόχρονα να απαντούν και σε όλες τις εισερχόμενες αιτήσει για έρευνα. Και βλέπετε στα στοιχεία, μιλάμε για ε, χίλιες, ε, πάνω από 1.200 του 2012 αιτήσει. Αυτό σημαίνει, αν το επιμερίσουμε, 10 αιτήματα την ημέρα. Άρα μια ερευνητική ομάδα έπρεπε να απαντά σε 10 αιτήματα την ημέρα πριν δημιουργήσουμε την ειδική μονάδα. στο ερώτημα που ετέθη ε, για τις ε, καταγγελίες που έρχονται από τις κρατικές αρχές και από τους ιδιώτες, το ερώτημα του κ. Σόντερκαρτ, αυτά τα στοιχεία εγώ τα βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Δυστυχώς δεν τα έχουμε για τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά ξεκινάμε και από εδώ και πέρα, από εδώ και στο εξής θα τα έχουμε. Μας προβλημάτισαν και εμάς Και εμάς μας εξέπληξαν. Δύο στοιχεία πρέπει να συγκρατήσουμε πιστεύω. Όσον αφορά τους ιδιώτες, ο Όλαφ είναι γνωστός ή όχι. Με εκπλήσει σε ορισμένα κράτη-μέλη και θα ονοματίσω ένα, τη Βουλγαρία για παράδειγμα, είναι πολύ γνωστό ο Όλαφ. Με έχει γίνει από τα μέσα μαζική ενημέρωση. Μέρ με ρωτήσετε γιατί, αλλά όλοι τον έμαθαν. οποτεδήποτε ο Όλαφ είναι γνωστός, αυτό ε, έχει ως αποτέλεσμα να απευθύνονται οι ιδιώτες στον Όλαφ. Σε άλλα κράτη-μέλη, όπως το δικό σας, κανείς δεν ξέρει τι είναι ο Όλαφ. Σχεδόν κανείς. Αυτό επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά επίσης ε, έχει σημασία και το ποια είναι η δημόσια εικόνα του Όλαφ κάτι που εξαρτάται από τις έρευνες που διεξάγει. Και όσον αφορά τις κρατικές αρχές, αυτές οι μεγάλες διαφορές που διαπιστώνουμε ε, σε σχέση με την συνεργασία του Όλαφ με τις κρατικές αρχές, νομίζω ότι όλα εξαρτώνται από την εμπειρία αυτής της ε, κάθε δημόσιας διοίκησης. Όταν ο Όλαφ έχει συνεργαστεί ικανοποιητικά με την αστυνομία, με την εισαγγελία, με τις διοικητικές αρχές ενός κράτους μέλους, αρχίζει να υπάρχει μια μεγαλύτερη ροή υποθέσεων. Δεν θέλω να κατηγορήσω τα κράτη-μέλη που δεν μας αποστέλουν ε, καταγγελίες. Μπορεί απλώς αυτό να σημαίνει ότι καταφέρνουν μόνα τους να αντιμετωπίζουν τις υποθέσεις απάτης που έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στον ε, προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθώ να είμαι πολύ αυτό που λέω. Μπορεί απλώς και μόνο να σημαίνει ότι οι εθνικές αρχές καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα χωρίς τη βοήθεια του Όλαφ. Κανείς δεν έχει το αλάθητο και δεν έχουμε έρθει εδώ να ζητήσουμε να ε, λαμβάνουμε περισσότερες καταγγελίες. Ήδη διαπιστώνεται ότι είναι δύσκολο να λαμβάνουμε, αλλά φαίνεται από τα στατιστικά στοιχεία ότι υπάρχει μια διαφορά, μια αναντιστοιχία μεταξύ των καταγγελιών που λαμβάνουμε από τις κρατικές αρχές και από τους ιδιώτες. Σε γενικές γραμμές πρέπει να πούμε ότι οι καταγγελίες που έρχονται από τις κρατικές αρχές είναι καλύτερα τεκμηριωμένες, είναι πιο ουσιαστικές. Μερικές φορές αυτές οι καταγγελίες που έρχονται από τους ιδιώτες ε, δεν ε, είναι τεκμηριωμένες, δεν βοηθούν, δεν έχει νόημα να ερευνηθούν. Τέλος, με ρωτήσατε ποιοι ερευνούν τις καταγγελίες, ποιος, ποιος διεξάγει τις έρευνες στον Όλαφ. Ναι, προφανώς το προσωπικό, το μόνιμο προσωπικό της υπηρεσίας, που είναι προσωπικό της Επιτροπής. Έχουμε επίσης ε, ε, έκτακτους ε, υπαλλήλους. Κάποιοι από αυτούς έχουν συμβόλαιο αερίστου χρόνου και κάποιοι ορισμένες συμβόλαιο ορισμένες διάρκειας. αλλά πρόκειται για ε, άτομα που είναι μέλη ε, του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του προσωπικού του Όλαφ. Επίσης υπάρχουν οι αποσπασμένοι από τα εθνικά κράτη-μέλη. Δεν είναι πολλοί, αλλά ε, μας βοηθούν και αυτοί σε ορισμένες έρευνες. Ορισμένοι επαγγελματικοί κλάδοι όπως για παράδειγμα οι εισαγγελείς, είναι πολύ δύσκολο να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες του Όλαφ ως μέλη του προσωπικού. Γιατί ε, χρειάζεται να γίνει ένας κατάλληλος διαγωνισμός. Δεν θα ήταν σκόπιμο να κάνει κανείς έναν διαγωνισμό ή να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έναν ε, διαγωνισμό στο επίπεδο του ε, υπαλλήλου AD5 και στο οποίο θα συμμετάσχουν δεκάδες χιλιάδες υποψήφοι ελείπουν στο προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δυσέβρετη γιατί γι' αυτό το προσωπικό το οποίο χρειάζεται σε περιορισμένο αριθμό θα πρέπει να το βρείτε με το να έχετε αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμενους. Πού βλέπετε τους εξωτερικούς ε, ε, υπαλλήλου. Είναι οι κρατικοί αποσπασμένοι. Α, το λέει η έκθεση. Η κυρία Γιάλα Σέντερ χωρίς μικρόφωνο. Έχουμε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Είναι οι λεγόμενοι ε, προσλαμβανόμενοι με σύμβαση ίντραμούρος, ενδοτυχικοί υπάλληλοι όπως τους λέμε. Έχουμε κάποιες εξωτερικές εταιρείες οι οποίες μας δίνουν υπηρεσίες αλλά μας δίνουν και προσωπικό για να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρα σε αυτές τις υπηρεσίες και αυτά τα άτομα τα οποία δεν ανήκουν στην Όλαφ δουλεύουν με την Όλαφ αλλά δεν αγγίζουν τις έρευνες καθόλου. Το ερευνητικό κομμάτι της Όλαφ δεν το δεν συμμετέχουν. Κατά τα άλλα, αν δεν, είμαι, αν δεν ήμουν απόλυτα σαφής, παραμένω στην διάθεσή σας. Και όποτε θέλετε, μια μέρα, κάποια μέρα, κάποτε, θα ήθελα να υποδεχτώ και την Επιτροπή σας στις εγκαταστάσεις της Όλαφ για μισή μέρα αν θέλετε να συναντήσει την ε, διοικητική ιεραρχία της Όλαφ, το προσωπικό και να δείτε επιτοπίως πώς εργαζόμαστε μέρα, μέρα και νύχτα, νύχτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Φιντά. Θα βγάλουμε ειστήριο με επιστροφή. Έχουμε γύρω στα 7 λεπτά. Η κυρία Γκρέσλε ήθελε να κάνει κάποιες παραπάνω ερωτήσεις. 7 λεπτά και μετά πρέπει να πάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ε, με συγχωρείτε κύριε Γενική Διευθυντά, αλλά με αυτά τα οποία λέτε για την έκθεση του 2012 και τα καλύτερα αποτελέσματα και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, εγώ βλέπω τα αντίθετα. Τα νούμερα του 2012 έχουν επηρεαστεί από την απόφασή σας να ανοίξετε σε μία μέρα 423 υποθέσεις από τις οποίες κλείσατε μετά τις μισές. Χωρίς αυτό θα είχαμε τελείως διαφορετικά νούμερα και το ξέρουμε και οι δύο. Επίσης τα υπόλοιπα ε, ε, λέτε μειώθηκε η διάρκεια της αξιολόγησης. Μα αν έχουμε 400 υποθέσεις που τις ανοίγουμε και τις κλείνουμε αμέσω, ε, ναι και εδώ πέρα αυτό επηρεάζει τη στατιστική έτσι. Δεν είναι άρα τόσο έγκυρα τα στοιχεία σας και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Το θέμα είναι αν έγιναν όλα αυτά σωστά. Το ζήτημα λοιπόν είναι ε, εάν ε, υπάρχει το ποσοστό σφάλματος. Το ποσοστό σφάλματος είναι 50%. 50% είναι τραγικό. Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι ποτέ δεν ήταν τόσο άσχημα προστατευμένα τα οικονομικά συμφέροντα της κοινότητας. Ανησυχώ πάρα πολύ. Σοβαρά μιλάω. Δηλαδή τόσο υψηλό ποσοστό σφάλματος είναι τραγικό. Μην με παρεξηγείτε προσπάθησα να δω τα νούμερα στην περίπτωση ε, για να δούμε ακριβώς και το ζήλο του Όλαφ. Δεν είναι δυνατόν σε μία στις 20 περιπτώσεις να μην συμβαίνει ακριβώς τίποτα. Όταν ξέρουμε πως υπάρχουν περιπτώσεις όπου επί σειρά ετών υπάλληλοι περιμένουν ο Όλαφ να ασχοληθεί με την υπόθεσή τους. Ξέρουμε και οι δύο Έχουμε και μία σχετική ακρόαση για το τι γίνεται δηλαδή με τους ε, ενδιαφερόμενους. Μιλάμε για ανθρώπινες καταστροφές εδώ πέρα, για ανθρώπινες τραγωδίες. Για την δε έκθεση του, την απαλλαγή του 2012 την ε, ψηφίσαμε προχτές. Το σύστημα λοιπόν που μας απασχολεί είναι το ε, σημείο υπαριθμών 66 που αφορά επίσης ε, και την ε, καταγραφή των τηλεφωνημάτων. Σας ευχαριστώ, κυρία Σέντερ. Ε, τηλεγραφικά, αλλά ο κύριος Κέστερ δεν απάντησε στο ερώτημα αυτό για τις υποθέσεις που εκκρεμούν εναντίον της ΟΛΑΦ και εναντίον του προσωπικού της ΟΛΑΦ. ποιε είναι αυτές οι υποθέσει αν μπορεί να, μας, να αναφερθεί σε αυτέ που υπάρχει αυτή τη στιγμή μετά από δράση τη Όλαφ, ανοιχτή δικαστική διαδικασία. Πέντε λεπτά κύριε Γενικέ. Υπέρμετρα πολλά τα πέντε λεπτά. Ελπίζω. δεν ε, διαχωρίσαμε απαντών στο τελευταίο ερώτημα. Δεν διαχωρίσαμε τις συνεχιζόμενες ερεύνες της Όλαφ επί τη βάση φορέως ή ιδρύματος. Ήταν κατανοημένες σε ό,τι αφορά τα μέλη των ευρωπαϊκών ε, οργάνων, το προσωπικό των ευρωπαϊκών οργάνων και σε λοιπά θέματα. Αλλά αν δείτε τις στατιστικές για μεμονωμένα θεσμικά όργανα, 10 για την Κομισιόν, 15 για το Κοινοβούλιο, πουχού. Και μετά έχουμε πιο κούτσικα θεσμικά όργανα, Eurojust, Europol, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και μια πληθωρική πολυμορφία αποκεντρωμένων φορέων όπου και εκεί είναι καθήκον μας να κάνουμε έρευνες και καμιά φορά το κάνουμε για την δουλειά μας τότε επειδή είναι μικροί αριθμοί θα ότι γίνονται έρευνες εν εξελίξη ή άρτη περατοτήσεις εξελίξεις και τότε θα μας επέκριναν ίσως και το Κοινοβούλιο το, για το γεγονό ότι υπάρχει μια έρευνα η οποία είναι εν εξελίξη για κάποιο αποκεντρωμένο φορέα ή για κάποιο συγκεκριμένο άτομο στο προσωπικό ενό οργάνου, ενό φορέα. Γι' αυτό δεν δώσαμε του αριθμού αυτού στην δημοσιότητα. Δεν με καταλάβατε πολύ καλά ή εγώ δεν εξήγησα τον την άποψή μου πολύ καλά. Έλεγα για τις περιπτώσεις τις οποίες εκλήθη η ΟΛΑΦ έναντι των δικαστηρίων όχι τις υποθέσεις που φέρατε εσείς στα δικαστήρια, πόσες φορές υπήρξε δικαστική ενέργεια κατά της ΟΛΑΦ που ζητήθηκε να καταθέσει η ΟΛΑΦ σε ε, εθνικά δικαστήρια ή στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αν υπάρχουν τέτοιε περιπτώσει κτλ. Α, τώρα το πιασα. Συγγνώμη. Συγγνώμη για την παρεξήγηση, κυρία αλλά Δεν τα έχω τα στοιχεία αυτά αλλά για το 2012 μας φέρανε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο Λουξεμβούργο σε μια διαδικασία κατεπήγοντος. Αντέδρασε μέσα σε βδομάδες ή σε μήνες στο δικαστήριο σε σχέση με μια συνεχιζόμενη έρευνα για μέλος του προσωπικού ενός θεσμικού οργάνου. Ναι, θα μπορούσα ακόμα και να σας πω ποιο ήταν, γιατί είχε δει τις εφημερίδες και έτσι αλλιώς οι αποφάσεις του δικαστηρίου δεν είναι δημόσιες. Τότε όμως ήταν συνεχιζόμενη η έρευνα για κάποιο μέλος του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου και πρόκειτο για τρία ή τέσσερα άτομα τα οποία είχαν προσφύγει εναντίον της ΟΛΑΦ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όχι μόνο ανεγνώρισε την πλήρη θεμητονομιμότητα των ερευνητικών μας δράσεων, αλλά περαιτέρω κατεδίκασε τα άτομα αυτά στην καταβολή των δικαστικών εξόδων. Αυτή είναι η μοναδική τέτοιου είδους υπόθεση το 2012. Αν δούμε τις στατιστικές τα τελευταία χρόνια, δεν είναι κάτι που γίνεται κάθε μέρα, αλλά είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Μπορεί οποιοδήποτε να προσφύγει αν εμπλέκεται κατά του της ΟΛΑΦ. Η τελευταία φορά που κάποιες πράξεις της ΟΛΑΦ θεωρήθηκαν ότι παραβιάζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία ήταν σε μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το 2008 που αφορούσε ακόμα παλαιότερες έρευνες της ΟΛΑΤ. Έκτοτε μπορώ να σας πω με απόλυτη ασφάλεια ότι ποτέ δεν θεωρήθηκε ότι έσφαλε η Όλαφ ή ότι παρεβίασε κάποια νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια έχει σταθεί σε δικαστικές διαδικασίες, αλλά μετά το 2008 ποτέ δεν θεωρήθηκε ότι έκανε κάτι κακό η Όλαφ. Κύριε Γκρέσλε, τι να σας πω τώρα σε εσά. Οι πυραμίδες χωρίς τις 19 περιπτώσεις που δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε να βάλουμε στις 419, οι ανοιχτές περιπτώσεις ε, πέρσι ήταν περισσότερες από τα προηγούμενα χρόνια. Και η διάρκεια των ε, ερευνών έχει βραχυνθεί και είναι ακόμα πιο σύντομη το 2013. Το βλέπετε αυτό στην τελική έκθεση, αλλά εμείς θα παρακολουθούμε μήνα με το μήνα. Αυτό δείχνει ότι μειώνεται η διάρκεια <clears throat> των ερευνών. Αυτό δεν είναι το αποτέλεσμα των διαβόητων 419 υποθέσεων που φέραμε από τα συρτάρια μας και ανασύραμε από τα χρονοτούλαπά μας. Αλλά είναι κάτι το οποίο οφείλεται στην αφοσίωση του θαυμάσιου προσωπικού που έχει η Όλαφ. Γιατί αυτά συνάδουν και με την στατιστική του εφετινού έτους όταν δεν υπάρχουν αυτές τις 419 υποθέσεις στις οποίες αναφέρεσαι. Εντάξει, εντάξει. Να είσαστε σίγουροι ότι θα δώσουμε πάντα στους εμπλεκόμενους τη δυνατότητα να σχολιάσουν το κάνουμε πάντα σε σχέση με τα θέματα αυτά και φυσικά με τον νέο κανονισμό από την 1η Οκτωβρίου θα έχουμε μια νομική υποχρέωση. Το κάνουμε, το κάνουμε όμως ήδη από την 1η Φεβρουαρίου με τρόπο ο οποίος είναι συνεπής και συνακτικός. Εγγράφος, εγγράφος. Μέσα στα πλαίσια της γραπτής διαδικασίας υπάρχει και μια ιστοσελίδα και υπάρχει και μια ενκύκλιος που δίδει εντολές στο προσωπικό της Όλαφ. Ετέθησε εφαρμογή με δική μου πρωτοβουλία στην 1η Φεβρουαρίου, ώστε πρωτού κλείσει η έρευνα θα πρέπει να έχει δυνατότητα ο εμπλακόμενος να είναι πληροφορημένος για την κατηγορία, δεν είναι ακριβώς κατηγορία, για το περιεχόμενο της υπόθεσης λοιπόν που τον εμπλέκει και δεύτερον να έχει τη δυνατότητα να δώσει προφορικά ή ενεγάφως να εκφράσει τις απόψεις του και να κάνει μια δήλωση. Αυτό γίνεται με συνεπή τρόπο από το Φεβρουάριο του 2012, ακόμα και αν μέχρι αμεθαύριο δεν αποτελεί αυτό μια νομική υποχρέωση. Εμείς προκαταλάβαμε τα αποτελέσματα του νέου κανονισμού. Στο παρελθόν, κυρία Γκρέσλε υπήρξαν κάποια μέλη του προσωπικού που δεν είχε γίνει συνέντευξη μαζί τους ή των οποίων η θέση είχε παραμείνει για πολύ καιρό υπό έρευνα αλλά όπως βλέπετε από τα στοιχεία αυτά αυτό δεν ξαναγίνεται πρώτον γιατί γίνεται συνέντευξη σε όλες τις περιπτώσεις ακόμα και αν δεν θεωρούμε ότι δεν δίνουμε συνέχεια σε αυτήν την υπόθεση και δεύτερον η διάρκεια των περιπτώσεων, ιδίω των περιπτώσεων όπου κάποιο άτομο πλήττεται από το γεγονός ότι είναι για πολύ μεγάλο διάστημα υπό εξέταση και μπορεί να θυγεί η ιεραρχική τους εξέλιξη. Γίνεται αυτό. Και στην περίπτωση Ντάλι κάνουμε κάθε προσπάθεια να δώσουμε προτεραιότητα στα θέματα αυτά για να μην αφήσουμε ξεκρέμαστη τη φήμη ενός ατόμου για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και κάναμε όλες τις απαραίτητες προσπάθειες και κάνουμε όλες τις απαραίτητες προσπάθειες ώστε το άτομο αυτό να έχει όλη τη δυνατότητα να εκφράσει την απόψη του ίσως υπερβολικά αλλά δεν μετανιώνω για τίποτα να εκφράσουν τις απόψεις τους για όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Σας ε, παρακαλώ να σταματήσετε γιατί έχουμε ξεπεράσει το πρόγραμμα κατά μισή ώρα. Με πάση περιπτώσει σας ευχαριστούμε κύριε Γενική Διευθυντά για την παρουσία σας για αυτά τα οποία μας είπατε, για τη συζήτηση, αλλά θα σας παρακαλέσω να σημειώσετε το εξής. Η Επιτροπή μας δεν θα επαναχωρήσει όσον αφορά τις γενικές αρχές της. Όσον αφορά τις απάτες, το θέμα της αποτελεσματικότητας των ερευνών θα τίθεται πάντα. Η αποτελεσματικότητα σημαίνει πόσες περιπτώσεις ερευνήθηκαν, πόσο καιρός χρειάζεται να ερευνηθούν, το ποσοστό σφάλματος ε, στο δυνατόν χαμηλότερο και γενικά βλέπουμε πως ε, ζητάμε παντού οικονομίες. Δεν κάνουμε οικονομίες από τον Όλαφ, γιατί θέλουμε, έχουμε το εξή όνειρο, ότι θα υπάρχει ένας Όλαφ, ε, ο οποίος κοστίζει, αλλά δεν υπάρχουν ε, απάτες, ε, δωροδοκίες και <laughs> οι πολίτες είναι άγγελοι. Και θα υπάρχεται απλά ως ένα είδος πυροσβεστικής. Αυτός είναι ο στόχος μας λοιπόν. Οπότε θα είμαστε απαιτητικοί Έρχεστε εδώ ξανά και ξανά και μια επίσκεψη και στην υπηρεσία σας δεν είναι κακή ιδέα. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο μέρος της ε, συνεδρίασης ε, και κλεισμένων των θυρών. Κύριε Στάς, νομίζω μπορείτε να έρθετε να αναλάβετε την προεδρία. thank you very